Chers Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ε, έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Για την ημερήσια λοιπόν ε, ε, διάταξη θέλω να προτείνω μια τροποποίηση μετά από το αίτημα της κυρίας Γκαρδιαθάβαλ να μας παρουσιάσει την έκθεσή της χρηματοδότηση για την ισότητα των φύλων αμέσως μετά τις ανακοινώσεις που θα κάνω τώρα. Εάν δεν σας δημιουργεί πρόβλημα, τροποποιούμε έτσι την ημερήσια διάταξη. Σήμερα το πρωί συνεδρίασαν οι συντονιστές και όρισαν οι συγητές για το θέμα ε, δημοσιονομικοί κανόνες για το γενικό προϋπολογισμό θα είναι η συγγήτριά μας η κυρία Γκρέσλε που είναι η μόνιμη η συγγήτρια της Επιτροπής Προϋπολογισμών και επειδή είναι συναρμοδιότητα με την Κοντ η Κοντ λοιπόν έχει ορίσει τον κύριο Ρίτσορντ Ashworth ως συνεισηγητή. Επίσης ορίσαμε εισηγητή για το θέμα οι μελλοντικέ προοπτικές για τεχνική βοήθεια στην πολιτική συνοχή και θα την αναλάβω εγώ. Η έκθεση αυξανόμενη συμμετοχή των, εταιρικών, των εταίρων στα διαθροτικά ταμεία είναι γνωμοδότηση θα την αναλάβει το ΕΛΚ. η Επιτροπή μας θα πρέπει να εκφραστεί επί των τριών μέσων που αφορούν το σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων θα το αναλάβει η σοσιαλιστική ομάδα μάλλον θα αναλάβει η σοσιαλιστική ομάδα την έκθεση για το Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συναρμοδιότητα με την ΤΕΒ. και τις άλλε δύο εκθέσεις για τα άλλα δύο μέσα. Λοιπόν θα τι αναλάβει η κυρία Γκαρδιαθάβαλ. Όσον αφορά τις επιπτώσεις της αποχώρηση της κυρίας Γεωργίευα που ήταν ε, επιφορτισμένη με τον προϋπολογισμό και το προσωπικό τίθεται το θέμα της ακρόασης για, την, για τον ή την διάδοχό της θα μας απασχολήσει μετά τη λήξη της διαδικασίας του προπολογισμού για τις αποστολές και τις αντιπροσωπείες και τις ακρόασεις για το 2017 υπήρξε μια τροποποίηση του προγράμματος αποστολών προβλέπουμε να πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία τέλη Ιουλίου κατά την Πράσινη Εβδομάδα αλλά την εποχή εκείνη το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο δεν συνεδριάζει. Οπότε αυτή η αποστολή θα γίνει το Μάιο. Ενώ η αποστολή για την Παλαιστίνη το Μάιο θα γίνει λοιπόν τον Ιούλιο. Αποφασίσαμε να προσθέσουμε μία ακρόαση για τις επιπτώσεις του Brexit. η διακοινοβουλευτική ομάδα θα γίνει την 31η Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου 17 και αποφασίσαμε για την Ολομέλεια να προτείνουμε ήδη πόροι μετά την έκθεση Μόντι που ε, θα έχει μέχρι τότε δημοσιευθεί και για τα εργαστήρια όπως τα λέμε γιατί όπως ξέρετε συνεργανώνεται αυτή η εκδήλωση EMPL Η Επιτροπή μας θα έχει ένα ειδικό εργαστήριο για την εκτέλεση του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου όπου θα συζητήσουμε την καθυστέρηση δέσμευσης και έναρξη των προγραμμάτων και θα επιδιώξουμε απλουστεύσεις μετά και το πρόγραμμα Omnibus. Τέλος όσον αφορά την αμοιβή για το συμβόλαιο με τον κύριο Κίραν Μπράντλεϊ ως ειδικού συμβούλου δεν θα γίνει ανταλλαγή απόψε με βάση το άρθρο 123 του ε, του κώδικου άλλους υπαλλήλου της Ένωσης. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Οπότε τώρα να δώσω το λόγο στη κυρία Γουαρδιαθάβαλ για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της για την ενωσική χρηματοδότηση για την ισότητα των φίλων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη για την αίτησή μου για αλλαγή την τελευταία στιγμή της ημερήσιας διάταξης, αλλά δυστυχώς πρέπει να απουσιάσω λίγο από τη συνεδρίαση για να πάω σε άλλη συνεδρίαση. Επομένως ήθελα να είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσω να κάνω την παρουσίαση της νομοδότησης ε, σήμερα και σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την αλλαγή. Όπως ε, πολύ σωστά είπατε, πρόκειται για γνωμοδότηση για τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται πλήρως σε θέματα ισότητας φύλων και στις αξίες της και στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται αυτή η προσπάθεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων, τα τελευταία χρόνια αυτή η αλλαγή και αυτή η όφηση δεν ε, ήταν όσοι θα έπρεπε. Και για παράδειγμα στην τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που γίνεται μια σύγκριση για το μισθολογικό χάσμα, διαπιστώνουμε από το 2008 όχι μόνο δεν βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά μάλλον υποχώρησε και λίγο. Και αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, θα χρειαστούν 118 χρόνια προκειμένου να εξαλειφθεί αυτό το χάσμα μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Προσφάτως, την ε, προηγούμενη εβδομάδα, πήγα στην Ισλανδία ε, και ε, μάλλον συγγνώμη, στην Ισλανδία έγινε είδηση το γεγονός ότι στο 8ωρο εργασίας οι γυναίκες από τις 38 ώρες, τις 14 τις δούλευαν δωρεάν γιατί ε, υπάρχει ε, διαφορά και έτσι οι γυναίκες έκαναν μια άτυπη απεργία και αποφάσισαν ότι από τις δύο και μετά θα φύγουν από τη δουλειά για να δείξουν ότι στην πραγματικότητα δουλεύουν δωρεάν από τις δύο και μετά και δεν θα ε, το ανεχτούν αυτό. Δεν συζητούμε όμως μόνο... Παρακαλώ. Και τι ώρα ξεκινούν τη δουλειά του, λέει ο πρόεδρο. Ό,τι ώρα και οι άνδρε. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά από τι δύο και μετά είναι δωρεάν όσοι δουλειά προσφέρουν. Μα εγώ είχα καταλάβει ότι από τη Δευτέρα το απόγευμα 7 Νοεμβρίου οι γυναίκες δεν πληρώνονται. Ε, είναι λίγο διαφορετικός τρόπος να δούμε το ίδιο πράγμα, αλλά ακόμα και αν θα έπρεπε να το κάνουμε, για να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα αυτό, ε, μέσω ε, διαπραγμάτευση για τον προπολογισμό δεν ε, ε, γίνεται να το κάνουμε. Ο πρόεδρος λέει ότι οι γυναίκε από τη Δευτέρα το απόγευμα στι 7 Νοεμβρίου μάλλον εργάζονται δωρεάν. Τέλος πάντων, δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για αυτό το χάσμα μεταξύ των μισθών, αλλά βλέπουμε και τι διαφορετική μεταχείριση υπάρχει για τις γυναίκες. Είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά όχι μόνο δικαιοσύνης, είναι θέμα και οικονομικής και ανταγωνιστικής δικαιοσύνης. Υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη του Eurofam, 170 δις εκατομμύρια είναι η ευρώ είναι η απώλεια ε, πρόκειται για δύο προπολογισμού τη Ένωση, άμα το δείτε, ε, για την προσπάθεια που γίνεται, αν κάνετε σύγκριση των στοιχείων που έχουμε. Και ε, πολλοί λοιπόν ε, διεθνείς οργανισμοί λένε ότι πρέπει να γίνει προϋπολογισμός ακριβώς για τα θέματα φύλου ώστε να μπορέσουμε ε, να μειώσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και τα χάσματα που υπάρχουν. Στον 21ο αιώνα φαίνεται ψέμα να λέμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν θα πω άλλα εισαγωγικά, θα ήθελα να το θέσω λίγο στο πλαίσιο. ξέρουμε βέβαια ποιε είναι οι διαφορές, αλλά θα δούμε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών γυναικών. Για να μείνω στα τη γνωμοδότηση και το τι μπορούμε να ζητήσουμε εμεί από πλευρά Επιτροπή Προπολογισμών στη γνωμοδότησή μα, ζητώ οι γραμμέ προπολογισμού να διευκρινίσουν σαφέστατα ποιοι είναι οι στόχοι που αφορούν ε, τη σχέση των φύλων και ποιο τμήμα του προπολογισμού έχει διατεθεί για να επιτευθούν αυτοί οι στόχοι. Επίση, ζητώ τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν συγκεκριμένε δείκτε ε, φύλου για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη επιλογή των προγραμμάτων και να λαμβάνονται υπόψη αυτά όταν θα γίνεται παρακολούθηση και αξιολόγηση. Στο παρόν ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο έχουμε 6 170 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για τον ε, προπολογισμό για θέματα φύλων. Είναι πολύ καλό αυτό, αλλά ε, γνωρίζοντας πολύ καλά πως έχει κατάσταση πρέπει να αυξηθούν αυτά τα ποσά στο επόμενο πλαίσιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Επομένω, θα πρέπει να υπάρχει σαφή προπολογισμό σε θέματα φύλου σε όλο τον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων από το 2020 και μετά. Μέχρι τούδε υπήρξε κάποια πολιτική βούληση να δούμε τα θέματα ισότητας φύλων μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά η γήκενη η ώρα αυτή η πολιτική βούληση να μεταφραστεί και σε συγκεκριμένα στοιχεία και εδώ όσον αφορά εμάς σε ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα κονδύλια για να μειωθούν αυτές οι ανισότητες. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Περιμένω σχόλια, τη συνεισφορά σας, τις παρατηρήσεις της, ώστε να έχουμε και μια γνωμοδότηση η οποία θα είναι πραγματικά χρήσιμη για να μειωθούν αυτές οι ανισότητες. Merci. Merci pour... Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ε, να ξεκινήσουμε την ανταλλαγή απόψεων. Η κυρία Μούντι. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την ε, Άιντα για την γνωμοδότησή της, για τη δική μου έκθεση στην Επιτροπή Γυναικών γράφεται αυτή η γνωμοδότηση, την χαιρετίζω. Πολύ συχνά η πόροι της Ένωσης είναι οι μόνη πόροι σε κάποια κράτη-μέλη που έχουν συγκεκριμένη αναφορά στα θέματα φύλου αλλά και γενικότερα στην Ένωση όπου λέμε πολύ ωραία λόγια, πολύ συχνά δεν ακολουθούνται από σωστά έργα. Γι' αυτό αυτή η γνωμοδότηση είναι ιδιαίτερα καλοδεχούμενη γιατί είναι και σαφέστατη και πολύ εξειδικευμένη. Προτείνει πολύ συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιτύχουμε σαφή αποτελέσματα που να ανταποκρίνονται στις προθέσεις μας που είναι να υπάρξει ισότητα των φύλων μέσω της χρήσης των ενωσιακών πόρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Νομίζω ότι η κυρία Μούντι εξέφρασε τα συναισθήματα όλων μας. Οπότε Εντάξει, είπατε κυρία Μούντι πολύ σωστά ότι πολλές φορές ε, τα λόγια απέχουν των έργων. Αυτό ισχύει βεβαίως ε, όχι μόνο για την ισότητα ανδρών γυναικών αλλά και για άλλα θέματα στην πολιτική για τον προϋπολογισμό τώρα του 17 πώς θα μεταφραστούν όλα αυτά θα μπορούσε ο κύριος Γιέντς Γκάια να μας πει τη γνώμη του. Πράγματι, κοιτάξτε, εκεί που πρέπει λιγάκι να προβληματιστούμε περαιτέρω είναι το πώς μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά ε, θέματα προπολογισμού με τη διάσταση του φύλου. Αυτό είναι ένα αίτημα του Κοινοβουλίου, επαναλαμβάνεται συνεχώ, σωστό είναι αυτό και εγώ συμφωνώ, αλλά και εγώ ως εισηγητής του προπολογισμού ε, ρωτώντας ε, σκέφτηκα το εξής ρώτησα τους συναδέλφους που γνωρίζουν καλά τα θέματα και τους είπα, μα εντάξει συγκεκριμένα τι ακριβώς θέλετε, τι ακριβώς σημαίνει η εγγραφή στον προβλογισμό της διάστασης του φύλου, δηλαδή σε σχέση με τους αριθμούς παραδείγματο χάρη. Οι αριθμοί οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν στο να επιτύχουμε τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Και πρέπει να σας πω ότι δεν έχω καταλήξει πουθενά. Γιατί το τι πρέπει να γίνει κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, ε, δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Σίγουρα μπορεί κανείς πολύ αφηρημένα να πει ότι απαιτούμε πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες. Ε, και τι είναι αυτό τι είναι αυτό σε συγκεκριμένου αριθμού, Και όταν το ρωτάω ε, πάλι πολύ συγκεκριμένα μου λένε ξέρετε κάτι, παραδείγματο χάρη στι ε, πόλει να χρησιμοποιούνται οι αστικέ συγκοινωνίε περισσότερο γιατί λιγότερε γυναίκε έχουν ε, αυτοκίνητα από ότι οι άντρε. Και κατ' ουσίαν όταν προάγει κανεί αστικέ συγκοινωνίε σε μια πόλη κατ' ουσίαν προάγει την ένταξη τη διάσταση του φίλου στον ευρωπαϊκό, στον ενωσιακό Προπολογισμό. Αυτή είναι μια άποψη. Εγώ πιστεύω ότι ε, είναι μια ερώτηση που με απασχολεί πάρα πολύ και θα δούμε αργότερα μια μελέτη αυτής της Επιτροπής και θα δούμε ότι χρειάζονται ακόμα κάποιες προσπάθειες για να καταλήξουμε ενδεχομένως σε μια συγκεκριμένη μελέτη η οποία θα έχει συγκεντρώσει παραδείγματα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το ΩΣΑ γιατί ξέρετε κάτι, εγώ ευχαρίστω θα ήθελα όλα αυτά να τα εφαρμόσω στην πράξη αλλά μέχρι τώρα δεν έχω καταλάβει ακριβώς καλό το αίτημα αλλά δεν έχω καταλάβει πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη δεν έχω καταλήξει στο πώς αυτό το αίτημα αίτημα μπορεί να λάβει σάρκα και οστά ως ένα καθαρά πολιτικό αίτημα. Για τις αμοιβέ, για παράδειγμα, των συνεργατών μας. Ελπίζω ότι δεν γίνονται διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Ντεπρέ, που ήταν εισηγητής για τον προπολογισμό του 16. Δεν υπάρχει διάκριση. Έτσι δεν είναι ο κύριος Ντεπρέ. Θα υπάρχει σίγουρα, αλλά δεν είχα την εντολή, δεν είναι εντολή να κάνω έρευνα. Δεν σημειώθηκε πουθενά ως διάκριση κάτι. Νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμεθα το στόχο. Πλήρης ισότητα από κάθε άποψη για όλα τα θέματα που δεν έχουν να κάνουν με την αναπαραγωγική διαδικασία των είδους φυσικά. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με τους προσανατολισμούς που προτείνει η συγκητριά μας. Αλλά έχω δύο ερωτήσεις. Μία για να καταλάβω τους ορισμούς και μία επί της ουσίας. Ε, νόμιζα ότι δεν έπρεπε να μιλάμε πια για φύλλο, έτσι δεν λέμε σεξ, λέμε genre, gender, όχι σεξ. Ή είναι ένα θέμα μετάφρασης. Εδώ βλέπω να λέει κάτι για σεξ. Και στα γαλλικά λέει το κείμενο αναφέρεται στο σεξ και όχι στο genre. Πρέπει λοιπόν και το γαλλικό κείμενο να αναφέρει μία και μόνο λέξη. Δεν με ενοχλεί ο όρος σεξ στα γαλλικά, αλλά αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο όρος genre, πρέπει πιστεύω το κείμενο να είναι συνεπές. Τώρα επί της ουσίας. Στο σημείο 2 της γνωμοδότησης θέλετε να υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες και νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπε και ο γενικός μας συζητητής να υπάρχουν δείκτες αναφύλλω να εφαρμόζονται κατά την επιλογή, αποτίμηση και παρακολούθηση όλων των δράσεων. Όλων των δράσεων. Αλλά ξέρετε, οι δράσεις είναι πολύ ευρία έννοια. Αν πρέπει όταν καθορίζουμε τους στόχους και τα αποτελέσματα έχει έννοια αλλά για όλες τις φάσεις και για όλες τις δράσεις κοιτάξτε αν έχετε προγράμματα τώρα που έχουν πολλές δράσεις πολλές διαφορετικές δράσεις θα πρέπει να αναπτύξετε ειδικού αναφύλο δείκτες για κάθε δράση ή είναι απλώς θέμα ορολογίας γιατί αν δεν είναι, τότε νομίζω ότι επιβαρύνουμε γραφειοκρατικά δυσβάστακτα τη λειτουργία μας. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να αναδιατυπωθεί αυτό, για να είναι σαφές ότι οι στόχοι των προγραμμάτων μας βεβαίω πρέπει να περιέχουν δείκτες για αυτά τα θέματα, ότι μετά την εκτέλεση να δούμε αν πραγματικά έγιναν σεβαστοί αυτοί οι δείκτες, αλλά για όλες τις δράσεις και όλες τις φάσεις, εδώ νομίζω ότι το παρακάνουμε. Πρόεδρος. Κυρία Καρδιά πραγματικά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Για τους στόχους όλοι συμφωνούμε. Και όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Εάν σε όλες τις προκηρύξεις όμως, γιατί ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό κάνει κάθε μέρα. Ο προπολογισμό είναι αναδιανεμητικός και όλα γίνονται μέσω προκηρύξεων. Αν τώρα πρέπει να βάλουμε επιπλέον δείκτες, είναι ήδη απίστευτος λαβύρινθος οι προκηρύξεις μας και όλα τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν αν χρειαστούν επιπλέον διαδικασίες, κάτι γενικότερο να πούμε. ούτω ώστε να είναι πιο κατανοητό τι πρέπει να κάνουν και όλοι όσοι παρακολουθούν. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι που θα περάσει την οτροπία όλων μα να ασχολούμαστε με την ισότητα των φίλων. Για να καταλήξει την κυρία Γαρδιαθάβαλ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα ζητήσει το λόγο για να απαντήσω στην συνάδελφο την κυρία Μούντι, γιατί σαφές ότι καταλάβαμε η μία την άλλη, αλλά μετά από τις επόμενες παρεμβάσεις οι άντρες φαίνεται ότι διατάρεξαν τα πάντα τελικά, λέει ο πρόεδρος. Ακριβώς, ναι, κυρία Γουαρδία Θαμπάλ. Ίσως θα μπορούσε να είναι και θέμα Ενημέρωση ή και πληροφοριών και εξηγήσεων. Το πρώτο σχόλιο που έκανε ο κύριο Ντεπρέ νομίζω ότι είναι θέμα μετάφρασης. Στο πρωτότυπο, το οποίο είναι γραμμένο στα αγγλικά, λέει gender specific. Επομένως, ε, δεν είναι ασήμαντο αυτό, διότι η ορολογία που χρησιμοποιεί κάθε χώρα ε, είναι πολύ σημαντική, πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε και να υπάρχει ομοιόμορφη ορολογία. Επομένω, το gender specific ή πολιτικέ φύλου, που θα μπορούσαμε να πούμε στα ισπανικά, είναι, τελείως, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά τους δείκτε σε όλες τι δράσει και σε όλα τα στάδια, δεν είναι σε κάθε δράση και σε κάθε σημείο και δεν θέλουμε ούτε να προσθέσουμε γραφειοκρατία ούτε να προσθέσουμε ελέγχου. Θέλουμε να υπάρχει ενημέρωση και να μπορούμε να θέσουμε κριτήρια στα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να λαμβάνουν υπόψη και τη μείωση αυτών των ανισοτήτων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα επιδοτούμενα προγράμματα ε, βάσει του προπολογισμού της Ένωσης υπάρχει πάντα μία αξιολόγηση για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και κανείς φυσικά δεν είναι αντίθετος, ε, φαντάζομαι, διότι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε μέσω του ευρωπαϊκού προπολογισμού είναι να υπάρχει προστιθέμενη αξία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τελείω δεν θα είχαμε ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ζητάμε το ίδιο και για το ε, θέμα των ε, πολιτικών του φύλου. Αν θέλουμε να έχουμε δείκτε που καταδεικνύουν ότι πηγαίνουμε να καλύψουμε αυτό το χάσμα ή τι ανισότητε, ε, πρέπει κάτι να κάνουμε γιατί αλλιώ δεν θα τα καταφέρουμε. Και αυτό λέω να έχουμε αξιολόγηση. Δεν λέω σε κάθε δράση και σε κάθε σημείο, αλλά τα προγράμματα πρέπει να έχουν σαφείς στόχου και οι στόχοι αυτοί να έχουν δείκτες και αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων να ε, ε, είναι για να δούμε αν πετυχαίνουμε αυτό που έχουμε καθορίσει ότι θα πετύχουμε. Χρειαζόμαστε αυτά τα κριτήρια και τους δείκτες γιατί αλλιώ δεν ξέρουμε αν πετυχαίνουμε του στόχου μα. Και ε, Ίσως δεν είναι η διατύπωση, γιατί βλέπω και τον κύριο Ντεπρέ που με κοιτάει αρκετά σαφής. Επομένω θα προσπαθήσω να την ε, διευκρινίσω. Κάνουμε ό,τι κάνουμε και με άλλες πολιτικές. Όταν κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές για την νεολαία, για παράδειγμα, ή για τους πρόσφυγες ή ευρωπαϊκές πολιτικές, πάντα ή θα ε, πρέπει να βάλουμε ή βάζουμε ε, αποτελέσματα, να έχουμε δείκτες οι οποίοι ε, θα αποδεικνύουν ότι πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό. Συμφωνούμε λοιπόν. Ναι, για τη συμφωνία αυτή θα ολοκληρώσουμε. Υπάρχει μια μελέτη η οποία ανατέθηκε σε κάποιο εξωτερικό συνεργάτη. Ε, περιμένουμε και τα συμπεράσματα βεβαίως, αλλά αν σκεφτούμε και τι δράσεις θα μπορούσαμε να έχουμε ε, στα πλαίσια αυτής της μελέτης, ε, θα μπορούσαμε να δούμε ότι τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Θα πρέπει λοιπόν να υποβάλλετε τροπολογίες μέχρι τις 14 Νοεμβρίου στις 12 η ώρα, ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών 8 Δεκεμβρίου και η επί Επιτροπή θα ψηφίσει στις 27 Ιανουαρίου η Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστούμε κυρία Θαμπάλη για αυτή την ε, γνωμοδότηση η οποία οδήγησε και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και στην οποία θα επανέλθουμε. Περνάμε τώρα στην ανακοίνωση που αφορά το κόστος ε, των υπόλοιπων φορέων που αφορούν στην κοινή αγορά ο κύριος Γκάιερ ήταν ε, υπεύθυνο για τη μελέτη αυτή και του δίνω το λόγο πριν ζητήσω από τον ε, εμπειρογνώμονα, τον οποίο καλωσορίζουμε, να μας παρουσιάσει τη μελέτη του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ξέρετε αυτές τις ημέρες έχω πάρα πολλές δουλειές, πολλά πράγματα που πρέπει να κάνω. Ως μόνιμος ηγητής για τους οργανισμούς εγώ έκρινα ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να προτείνουμε αυτή τη μελέτη. Και πρέπει να σας πω, χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι οι συντονιστές συμφώνησαν και αυτοί μαζί μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από πολλά χρόνια συντάχθηκε μία μελέτη που είχε τον τίτλο «Το κόστος της μη ύπαρξη Ευρώπης». Με άλλα λόγια δηλαδή, τι κόστος θα προέκυπτε αν καταργεί το η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί αναφέρεται ποιο θα ήταν το διοικητικό κόστος ε, το τι αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των κρατών μελών επρόκειται περίπου για 1.000 εκατομμύρια, ένα τρεις, ένα τρεις κατ' ουσίαν. Ένα τρεις ε, το οποίο ε, εξοικονομείται κυρίως μέσω του ότι ορισμένες διαδικασίες διεκπεραιώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν ήταν η κεντρική ιδέα. Η κεντρική ιδέα που οδήγησε στο να σκεφτούμε ας κάνουμε το ίδιο και για τους οργανισμούς. Τότε εγώ μόλις είχα μπει στην Επιτροπή Προπολογισμών με κάλεσα να μιλήσω στη γερμανική τηλεόραση και στο τέλος η συντονίστρια της συζήτηση με ρώτησε εσείς πού θέλετε να προβείτε σε εξοικονόμηση κονδυλίων. Και εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ε, τους είπα ότι ξέρετε κάτι δεν είναι τόσο εύκολο να κάνουμε εξοικονομή κονδύλιων ε, στον προεπλογισμό. Συνήθω ε, έχουμε πάρα πολύ καλέ ιδέε του που να επενδύσουμε κονδύλια, το που να περικόψουμε κονδύλια. Αυτό ε, δεν το ήξερα να το πω. Κάτι ψέλισε εκεί και στο τέλο της συνέντευξη τη ρώτησα ε, και εσεί τι υπονοούσατε, τι υπενηχθήκατε Και είπε η συγκεκριμένη Ίστια να σα πω κάτι όλοι αυτοί οι οργανισμοί που είναι υπερβολικά πολύ μα δεν του χρειαζόμαστε. Έκτοτε λοιπόν εγώ παρακολούθησα αυτό το θέμα στην εξέλιξή του, ε, το συζήτησα και το παρακολούθησα και σε σχέση με τους ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι θέλουν να καταργηθούν οργανισμοί και λένε «μα είναι πάρα πολύ». Αλλά εγώ δεν άκουσα κάτι πολύ συγκεκριμένο από αυτού. Δηλαδή σίγουρα καλό είναι να δούμε κατά πόσον όλοι αυτοί οι οργανισμοί πράγματι εκπληρώνουν το στόχο για τον οποίο έχουν συσταθεί. Αλλά ξέρετε σε τελική ανάλυση πιο σημαντικό είναι να εξακριβώσει κανείς κατά πόσον αυτή η δουλειά που διεκπεραιώνει οι οργανισμοί κατά πόσον αυτή σχετίζεται με ευρωπαϊκή υπεραξία. Και αυτό ήταν και ο στόχος της μελέτης. Δηλαδή, κάποιες ε, διαδικασίες ε, που διεκπεραιώνονται από τους οργανισμούς. Αν αυτές διεκπεραιώνονται ξαφνικά αυτές οι διαδικασίες από τα 28 κράτη-μέλη ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά πόσον το αποτέλεσμα θα είναι θετικό ή όχι. Η μελέτη είναι πολύ ενδιαφέρουσα και περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση των ε, αποτελεσμάτων της μελέτης. Ο κύριος Τζακ Μάλεν θα απαντήσει στην αδημονία του κύριου Γκάιερ να ακούσει. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης για το κόστος της κατάργησης, της μη ύπαρξης των οργανισμών σε σχέση με την εσωτερική αγορά. Τον οργανισμό που συνδέονται με εσωτερική αγορά. Είναι ακόμη προσωρινά τα αποτελέσματα. Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης της μελέτης. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο. Νομίζω ότι αναγράφεται στην έκθεσή μου ότι είναι προσωρινή έκδοση. Στα 15-20 λεπτά που έχω διάθεσή μου, θέλω να σας κάνω μία επισκόπηση των στόχων και της μεθοδολογίας, αλλά και των πορισμάτων της μελέτης. Οπότε, ποιοι ήταν οι στόχοι της μελέτης. Τέσσερις. Πρώτον, να εξετάσουμε την επίπτωση της ύπαρξης των οργανισμών στον ενωσιακό και τους εθνικούς προϋπολογισμούς και να εξετάσουμε εάν θα ήταν διαφορετική η επίπτωση εάν εφαρμόζαμε εναλλακτικές λύσεις για να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Να παρέχουμε δηλαδή τις ίδιες δραστηριότητε και υπηρεσίες σε εθνικό και όχι ενωσιακό επίπεδο. Και αυτό που συνδέεται είναι λοιπόν τα ωφέλη και το κόστος. Και τρίτον, εάν τα ωφέλη που προκύπτουν από την διατήρηση εναρμονισμένων κανόνων στα 28 κράτη-μέλη είναι αξιόλογα και ποια είναι η προστιθέμενη αξία για διάφορους βασικούς εμπλεκόμενους, τις εθνικές αρχές, αλλά και επιχειρήσεις, αλλά και διεθνείς οργανισμούς. Τι μελετήσαμε. Μελετήσαμε 7 τέτοιους οργανισμούς. Αναφέρονται εδώ. Είναι για τα διενωτικά δικαιώματα, ασφάλεια της αεροπορίας, φάρμακα, χημικές ουσίες και τρεις ε, οργανισμοί χρηματοπιστωτικής ε, επιτήρησης, ε, η ΕΣΜΑ, η Τραπεζική Αρχή και η Αρχή για τις ασφάλειες και τις επαγγελματικές συντάξεις. Η έρευνα που κάναμε κράτησε τους τελευταίους δύο-τρεις μήνες. Κάναμε πολλές συζητήσεις με τις ε, οργανώσεις αυτές, με εθνικές αρχές, επιχειρήσεις όπως η Airbus και ενώσεις όπως η Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Εταιριών και οργανισμών, φαρμακευτικών οργανισμών καλύτερα. Τώρα για τη μεθοδολογία. Το κόστος της μη Ευρώπης αναφέρεται. Οι μελέτες δηλαδή για το κόστος της μη Ευρώπης. Και αυτό που κάνουμε εμείς είναι διαφορετικό αν και εξετάζουμε το ίδιο θέμα, αλλά η μεθοδολογία μας είναι λίγο διαφορετική. Οι μελέτες για το κόστος της μη Ευρώπης εστιάζουν κυρίως, θεωρώ, στο κόστος της μη ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας. Ενώ η δική μας μελέτη είναι το κόστος της μη Ευρώπης που εξέταζε κάτι που ήδη υπάρχει, δηλαδή αυτές οι οργανώσεις, αυτοί οι φορείς, και προσπαθούσαμε να υπολογίσουμε τι θα συνέβαινε αν δεν είχαν υπάρξει. Είναι κάπως διαφορετική προοπτική. Η ουσία της μεθοδολογίας βασιζόταν στην εξέταση, τριών διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων. Πρώτον, αυτό που υπάρχει τώρα και το κόστος λοιπόν των 7 αυτών φορέων. Δεύτερον, η βέλτιστη περίπτωση ή ίσως θα έπρεπε να ε, περιγραφεί σαν η λιγότερο κακή εναλλακτική λύση, δηλαδή εάν τα καθήκοντα των φορέων αυτών τα ανελάμβαναν τα κράτη-μέλη, ενώ το ρυθμιστικό πλαίσιο σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα τα συστήματα αμοιβαίων αναγνωρίσεων παρέμεναν ενισχύ. Και η τρίτη, που ήταν η χειρότερη αναλλακτική λύση, θα ήταν εάν δεν υπήρχε τέτοιο ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί η αμοιβαία αναγνώριση ε, σιγά σιγά υποβαθμίζεται και τελικά καταραίει. Οπότε τα κράτη-μέλη θα έπρεπε το καθένα να έχει κάποιες παρόμοιες δομές και οι εταιρείε που θα στρέφονταν προς αυτούς τους οργανισμούς θα έπρεπε σε κάθε χώρα να πάνε σε διαφορετικό φορέα για να κατοχυρώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Λοιπόν, να δούμε τώρα τα τρία αυτά σενάρια, τις τρεις αυτές εναλλακτικές λύσεις. Κυρίως θα ασχοληθώ με το δεύτερο που είναι το πιο ενδιαφέρον. Τώρα, πώς έχει τώρα η κατάσταση η βάση αναφοράς δηλαδή. Εξετάσαμε 7 φορεί. Συνολικό προπολογισμό έχουν 1,112 δι. Που είναι το 13% του προπολογισμού όλων των οργανισμών. Αλλά ένα πολύ μικρό τμήμα προέρχεται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, Γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί διάφορες από αυτές τις ε, οργανώσεις, διάφοροι από αυτούς τους οργανισμούς χρηματοδοτούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ποσά τα οποία χρεώνουν τους χρήστες. Για παράδειγμα, ο Οργανισμός Διανοτικής ε, Ιδιοκτησίας και ο Οργανισμός Φαρμάκων γύρω στο 90% αν όχι παραπάνω από τον προπολογισμό τους είναι φορές από τον ιδιωτικό τομέα όταν θέλουν ακριβώ να πιστοποιήσουν υπηρεσίε και προϊόντα σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Ενώ όσον αφορά κάποιες, ε, ε, κάποιες, ε, κάποιους φορείς επιτήρησης, για παράδειγμα για την τραπεζική αρχή, το 2015 ο προϋπολογισμός της ήταν γύρω στα 30 εκατομμύρια, εκ των οποίων 40% περίπου ήταν από τον ενωσιακό προϋπολογισμό, αλλά συνολικά Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το κόστος των οργανισμών δεν φέρεται κυρίως από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Να δούμε τώρα τι θα συμβεί αν αλλάξει τίποτα. Έχοντας συζητήσει με αυτούς τους φορείς, θεωρούμε ότι οι πόροι τους οποίους ε, δαπανούν θα μειωθούν γιατί θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά του. Τα στατιστικά που μας έχουν δώσει, οι περισσότεροι φορεί είναι, ε, είναι ότι ο αριθμό των διαδικασιών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνία με τους οποίους ασχολούνται ε, αυξάνονται κατά 5 με 10% το χρόνο ενώ ο προπολογισμό τους μειώνεται. Κάποιοι οργανισμοί και ιδιαίτερα οι προπολογισμοί στον χρηματοπιστωτικό τομέα μπορεί να αυξηθούν, ενώ αλλού θα μειωθούν. Συνολικά όμως μειώνονται. Τώρα, το πρώτο από τα δύο εναλλακτικά σενάρια. Το σενάριο αυτό προβλέπει ότι θα συνεχιστεί να ισχύει το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά ότι οι λειτουργίες των ευρωπαϊκών φορέων θα αντικατασταθούν από εθνικούς φορείς. Αυτό θεωρούμε ότι σημαίνει επιπλέον κόστος 160 με 170 εκατομμύρια το χρόνο, εάν τα καθήκοντα των ευρωπαϊκών φορέων μεταφερθούν στα κράτη-μέλη. Και αυτό το επιπλέον κόστος θα προκύψει εν μέρη από την ανάγκη δημιουργίας νέων φορέων, νέων υπηρεσιών, που θα πρέπει να αναλάβουν πολύ περισσότερες λειτουργίες από αυτές που έχουν ήδη, στην περίπτωση που υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι φορείς. Βέβαια, δεν θα υπήρχε ισο, ισομερής κατανομή όλων αυτών των συμπληρωματικών στοιχείων κόστους σε όλες τις χώρες. Αν δεν υπήρχε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν ε, ε, εκτεταμένη αεροπορική βιομηχανία θα έπρεπε να αναλάβουν το κόστος ε, της παροχής αυτών των υπηρεσιών. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα το Γραφείο Διπλωμάτων Αριστεχνίας, σε αυτή την περίπτωση από ό,τι φαίνεται θα έπρεπε, εάν καταργεί το αυτό το γραφείο, τότε όλα τα κράτη-μέλη θα ανελάμβαναν περίπου ισομερό το κόστος. Οπότε Το τι θα πληρώσει το κάθε κράτος μέλος εξαρτάται από την έκταση ε, της αντίστοιχης δραστηριότητας σε κάθε κράτος μέλος. Τώρα το δεύτερο σενάριο. Όταν δηλαδή, εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι φορείς, αυτές οι υπηρεσίες, κάποια στιγμή στο μέλλον, το ρυθμιστικό πλαίσιο θα αρχίσει σιγά σιγά να καταραίει. Διότι θα υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο, θα μειώνεται όλο και περισσότερο η αμοιβαία αναγνώριση. Και τότε θεωρούμε ότι ιδιαίτερα για τους τέσσερις φορείς που έχουν να κάνουν με την ενιαία αγορά, οι επιχειρήσεις των κλάδων αυτών θα έπρεπε να καταχωρήσουν τα προϊόντα τους σε κάθε μία από τις χώρες. Και εδώ έχουμε λοιπόν αύξηση του κόστου γιατί οι εθνικές εισφορές, οι εθνικές αμοιβέ για καταχώρηση, άμα δούμε από χώρα σε χώρα πώς λειτουργούν, αν, αν πρέπει λοιπόν να πιστοποιήσεις τα προϊόντα σου σε όλες αυτές τις χώρες, θα υπάρχει συσσόρευση του κόστους, θα είναι πολύ περισσότερο το κόστος από το να έκανες μία μόνο πιστοποίηση έναντι ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Έχουμε συγκεντρώσει τα στοιχεία μας και θεωρούμε ότι αν ίσχυε το δεύτερο σενάριο, εάν οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να καταχωρήσουν τα προϊόντα τους σε πολλές χώρες, αυτό θα πρόσθεται γύρω στα 500 εκατομμύρια έως 1 δις στο κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό ποσό. Κατά πολύ υπερβαίνει τα μικρότερα ποσά των 160 εκατομμυρίων που μπορεί να χρειαζόταν να δαπανίσουν τα κράτη-μέλη για να επεκτείνουν τη λειτουργία των υπαρχόντων οργανισμών τους. Πέρα από τα στοιχεία που σας έδωσα, υπάρχουν και αφανή στοιχεία κόστους για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν είναι μόνο το ότι θα χρειαστεί να πληρώσουν επιπλέον το κόστος της καταχώρησης. Υπάρχει και το κόστος ε, υποβολής αιτήσεων σε πολλούς οργανισμούς, σε όλες τις χώρες Ευρώπης για να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους, για να διοδοτήσουν τα προϊόντα τους. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε και με τον χρόνο που είχαμε, δεν μπορούσαμε να εξετάσουμε όλα τα στοιχεία αναλυτικά, αλλά τα στοιχεία που μας έδωσαν διάφορες επιχειρήσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα ήταν υψηλό αυτό το κόστος, πολύ υψηλότερο. Και κάτι άλλο ο καθορισμός, ο ποσοτικός καθορισμός του κόστους της μη ύπαρξης φορέων είναι πολύ δύσκολο στην περίπτωση των φορέων ε, χρηματοοικονομικής επίβλεψης. Είναι πολύ δύσκολο να αναφέρουμε ένα ποσό για το ποιο είναι το οικονομικό όφελος από την ε, σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρώπη. Για όλους αυτούς τους οργανισμούς υπάρχουν ε, και άλλες δαπάνες που είναι δύσκολο να καθοριστούν εάν δεν υπήρχαν. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί βεβαίως έχουν μεγάλη πείρα, τεχνογνωσία, ο οργανισμός φαρμάκων έχει 4.500 εμπειρογνώμων στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί για νέα φάρμακα, έχουν βάσεις δεδομένων που περιέχουν ε, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και που είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμα από ότι αν έπρεπε να ρωτήσεις ε, βάσεις δεδομένων σε κάθε χώρα και είναι πολύ σημαντικός ο διεθνής ρόλος που παίζουν αυτοί οι φορείς για παράδειγμα στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας μας είπαν ότι θα επιστρέφαμε στη δεκαετία του 60 εάν καταργούσαμε αυτό το φορέα κάθε χώρα θα έπρεπε να έχει το δικό της σύστημα για να ε, αδειοδοτεί τα αεροσκάφη που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες και θα μπορεί να ήταν διαφορετικά τα κριτήρια και από πλευράς βέβαια των κατασκευαστών αεροσκαφών. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η, η πείρα. Εάν λοιπόν καταργηθούν αυτοί οι φορείς, θα υπήρχαν επιπτώσεις ε, για την τοπική οικονομία των περιοχών ε, όπου λειτουργούν. Όλες μαζί, όλοι μαζί οι 7 οργανισμοί έχουν 3.500 εργαζόμενους. Βέβαια κάποιες θέσεις εργασίας θα δημιουργούν το αλλού, μάλλον εδώ στις Βρυξέλλες, για να αναλάβουν τις λειτουργίες που δεν θα μπορούσαν πλέον να εκτελέσουν οι φορείς που δεν θα υπήρχαν. Οι οργανισμοί αυτοί επίση δίνουν σωστή πληροφόρηση που επιτρέπουν ε, καλύτερο σχεδιασμό της πολιτικής. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι φορείς, κάποιες από αυτές ε, τι υπηρεσίε προσφοράς συμβουλών και γνώσης στα ενωσιακά όργανα θα έπρεπε να μεταφερθούν εδώ στι Βρυξέλλε. Θα υπήρχε λοιπόν επίπτωση στην τοπική οικονομία και θα υπήρχαν και έμεσε απώλειε θέσεων εργασία από όλου ε, όσου ε, εργάζονται σε σχέση με του φορεί αυτού και του παρέχουν υπηρεσίε. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι φορεί και επανέρχονται εδώ, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιε λειτουργίε. Δεν πήγαινε στα κράτη-μέλη. Βέβαια, η Κομισιόν θα μπορούσε να προσλάβει και άλλου υπαλλήλου ή να επιφορτήσει του υπάρχοντε. Αλλά πιστεύω πω θα ήταν δύσκολο αυτό επειδή είμαστε σε κλίμα δημοσιονομικών περικοπών. Οπότε δεν θα ήταν τόσο ολοκληρωμένη και σαφής η παροχή συμβουλών για τη διαμόρφωση της πολιτικής. Τέλος. Τα γενικά απορίσματά μας, όπως σας είπα, είμαστε σε φάση ολοκλήρωσής τους. Αναμφίβολα, έχοντας εξετάσει το θέμα, θεωρούμε ότι το κόστος λειτουργίας αυτών των φορέων είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος που θα προέκυπτε εάν επανέρχονται στα κράτη-μέλη ή αν αναλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι λειτουργίες αυτές. Τώρα είναι δύσκολο βέβαια να καθορίσουμε ποια είναι η διαφορά του κόστους. Είναι δύσκολο να συγκρίνεις ε, την υπάρχουσα κατάσταση με μια υποθετική κατάσταση. Βέβαια θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε την εξέταση και σε άλλους φορείς θεωρούμε ότι αν θεωρείτε ότι είναι καλή δουλειά που κάνουμε μέχρι τώρα, θα ήταν σκόπιμο να εξετάσουμε το κόστος και το όφελος από τη λειτουργία και κάποιων άλλων φορέων που εργάζονται σε σχέση με την εσωτερική αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ρωτήσω τον κύριο Γκάγερ εάν ικανοποιήθηκε η ανυπομονησία του. Ε, πρέπει να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένο με την ε, έκθεση και με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι πράγματι μπορεί κανείς να καθορίσει ποσοτικά την εξοικονόμηση κονδυλίων σε σχέση με τους ε, οργανισμούς ε, και σε σχέση με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένες υπηρεσίες οι οποίες πράγματι είναι καλύτερα να προσφέρονται κεντρικά αντί μεμονωμένα στα 28 κράτη-μέλη. Και τα στοιχεία δεν είναι τόσο εντυπωσιακά για τους προϋπολογισμούς ή για τον ε, προεπλογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι ότι το κόστος το οποίο θα προέκυπτε από κάποιο συγκεκριμένο ε, τομέα της οικονομίας, το κόστος αυτό θα ήταν τεράστιο. Ακούσαμε για ένα δις παραδείγματο χάρη και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Θεωρώ λοιπόν ότι Πράγματι, ε, ε, αυτά όλα που ακούσαμε μας βοηθούν στο να αποκρισταλώσουμε πολιτικά την άποψή μας και αν τελικά ε, συζητηθούν λίγο περισσότερο σε βάθος όλα αυτά τα επιχειρήματα, τότε θα υπήρχε μεγαλύτερη αξιοπιστία αυτών των οργανισμών. Βεβαίω δεν ξέρω ε, κατά πόσον σε μια μελέτη μπορεί κανείς ε, να συσχετίσει οργανισμούς και με ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα. Αυτό που καθίσατε περισσότερο σαφέ είναι στον τομέα των αερομεταφορών και στον ε, φαρμακευτικό τομέα. Εκεί η υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι εταίροι για να μπορεί κανείς να ε, ενταχθεί στον αντίστοιχο οικονομικό κλάδο. Εκεί τα πράγματα είναι απόλυτα σαφείς. Ε, όταν πρόκειται για την λειτουργία αυτών των οργανισμών, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να υπενθυμίζει κανείς τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, τους αριθμούς. Εγώ θυμάμαι λιγάκι, έχω κάνει μια οδυνηρή εμπειρία στο θέμα της διαμόρφωσης των εισφορών. Δηλαδή είχε τεθεί το ερώτημα του κατά πόσο ενδεχομένω τα πλεονάσματα που προκύπτουν από τη λειτουργία των οργανισμών να μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει για τα δικά του αδικητικά έξοδα ή για τον νοσιακό προϋπολογισμό. Και μου είχε πει ή μάλλον έχω κατά νου ε, κάτι που ελέγχθη από εκπροσώπους αυτών των τομέα της αεροπλοείας ε, όταν εγώ ε, συνέντασα μια έκθεση για την ΝΑΖΑ και θα το πω έτσι με λίγα λόγια. Εκεί η εκπρόσωπος μου είχε πει ότι το ύψος της εισφοράς για μας δεν είναι τόσο σημαντικό. Σημαντικότερο είναι πόσο γρήγορα μπορεί να οργανιστεί ο οργανισμός και πόσο γρήγορα μπορεί ο οργανισμός να προσφέρει μια συγκεκριμένη υπηρεσία στον κλάδο. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πόσο γρήγορα μπορεί ο συγκεκριμένο οργανισμό να ε, εκδίδει πιστοποιητικά στην, στον τομέα της αεροπλοεία για να λειτουργεί καλύτερο ο αυτό. αυτός. περιπτώσει, εγώ θα τα δω λιγάκι, θα τα δω καλύτερα ε, όλα αυτά που αναφέρει η μελέτη και όσον αφορά στον ε, προϋπολογισμό αλλά και στον βασικό κανονισμό που θα προκύψει, σίγουρα θα πάρω ε, κάποια επιχειρήματα από τη μελέτη που ακούσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Σντεσόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τα αποτελέσματα του έργου των διαφόρων οργανισμών και είναι αδιαπραγμάτευτη η κριτική μας. Δεν αφήνουμε τίποτα όρθιο, ψάχνουμε τα πάντα και αξιολογούμε το έργο όλων των οργανισμών. Δεν λέμε απλώς ότι όλα ωραία και καλά. Πολύ συχνά έχουμε αρνηθεί να δώσουμε απαλλαγή σε κάποιον οργανισμό. Εγώ ήμουν ο μόνιμος ε, επιτροπή, ε, ε, εισηγητής του ΕΛΚ για τις διάφορους οργανισμούς και επισκέφθηκα 19 εξ αυτών. Έχω πάει σε όλη την Ευρώπη, έμεναν τουλάχιστον μισή ημέρα σε κάθε οργανισμό, εξέταζα πάρα πολύ προσεκτικά τη δουλειά τους, τα προβλήματά τους και αυτό έγινε στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Όπως και ο κύριος Γκάιερ, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να απαντήσω την ερώτηση για τους οργανισμούς. Οι οργανισμοί κάνουν καλή δουλειά και έχουν καλό προσωπικό, παρόλα αυτά όμως τους αξίζουν και κάποιες επικρίσεις και πρέπει να σκεφτούμε και κατά πόσον θέλουμε να συνεχίσουμε να τους στέλνουμε χρήματα. Ε, δεν ε, καταφέρνουν ε, να εξηγήσουν πολύ καλά το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και την προσπάθεια που καταβάλουν. Από αυτά που ακούσαμε από τον Τζακ Μάλεν, έχουμε μια μερική εικόνα, είναι μερική η μελέτη. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να δω και τα τελικά συμπεράσματα. Μην με παρεξηγείτε, ε, οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μια χαρά είναι. Αλλά αν είχαμε 28 διαφορετικούς ρυθμιστικούς φορείς που ε, θα έλεγχαν το κατά πόσον μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα, ε, καταλαβαίνετε τι θα συνέβαινε. Έχω πείρα από αυτά τα θέματα. Στην Τσεχική Δημοκρατία έχουμε μια χούφτα εμπειρογνώμονες ε, για την αεροπορία και νομίζω ότι δεν θα ήταν στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό πριν καν συζητήσουμε χώρες όπως η Κύπρος και η Μάλτα. Ε, δεν ε, θα ήθελα να με κατηγορήσετε βέβαια μόλις φύγω από την αίθουσα γιατί επικρίνω τις μικρότερες χώρες. Αυτό που λέω είναι ότι οι μικρές χώρες, ε, το Λουξεμβούργο, οι χώρες της Βαλτικής δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν τέτοιους εμπειρογνώμονες για να κάνουν αυτές τις διαδικασίες. θα ήθελα λοιπόν εγώ να μπορέσουμε να το ποσοτικοποιήσουμε αυτό και να υπολογίσουμε πόσο θα κόστιζε αν είχαμε 28 ξεχωριστούς οργανισμούς που θα έκανε αυτές τις δουλειέ. Ε, Παραδείγματο χάρη, πήγα στον Οργανισμό Ασφαλεία των Τροφίμων. Ε, Αυτέ οι ομάδε εκεί κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μπορούν να κάνουν ανταλλαγή πληροφοριών ε, ε, στο στο τσακ, πραγματικά. Είναι εξαιρετικό το πόσο γρήγορα γίνονται αυτά τα πράγματα. Εάν υπήρχαν 28 κράτη-μέλη που δούλευαν εκ παραλίλου, συζητούσαν το κατά πόσο θα πρέπει να απαγορεύσουμε αυτή την ουσία τώρα ή να το απαγορεύσουμε αύριο ή αν θα πρέπει να το κοιτάξουμε και από όλε τι πλευρέ το θέμα, ε, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Είμαι πολύ ε, Χαρούμενο που ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να αφιερώσουμε πολύ περισσότερο χρόνο σε αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να γίνει σύντομα μια νέα συζήτηση, διότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι οργανισμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν θησαυρό. Είναι ένα κόσμημα στα χέρια μα και δυστυχώ είναι βαθιά χωμένο κάτω από τη γη και δεν το βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Μαραγάγου. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη σας και τη χαιρετίζω. Αλλά ξεκινάει με μια βασική υπόθεση. Αναλύουμε τη λειτουργία των φορέων, θεωρώντας ως δεδομένο ότι η λειτουργία το περιεχόμενο της αρμοδιότητας, αν έχει έννοια, θεωρούμε ότι έχει έννοια να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι κράτους μέλους. Και εγώ είμαι πεισμένος ότι βεβαίως, βεβαίως ισχύει αυτή η προϋπόθεση. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να το εξηγήσουμε περισσότερο. Να εξηγήσουμε δηλαδή γιατί είναι καλύτερα να γίνεται σε ευρωπαϊκό και όχι εθνικό επίπεδο. και κατόπιν μπορούμε να δούμε και διάφορες άλλες εναλλακτικέ λύσεις. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πούμε ότι ναι πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά από την Κομισιόν, όχι από χωριστούς οργανισμούς. Πολλές από αυτές τις λειτουργίες δεν γίνονται στα κράτη-μέλη από κάποιο φορέα, αλλά από τη δημόσια δίκηση. Δεν λέω πως είναι η καλύτερη λύση, αλλά πρέπει να την εξετάσουμε. Ή άλλη δυνατότητα, κάποιοι τέτοιοι οργανισμοί για να κάνουμε οικονομίες κλίμακας, να θεωρηθεί ότι μπορούν να ενοποιηθούν στα πλαίσια κάποιας ενοποίησης ε, θεματολογικής. Γιατί εδώ ασχοληθήκαμε με 7, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες. Θα μπορούσαμε να τις ενοποιήσουμε για να επιτύχουμε περισσότερα αποτελέσματα εξοικονομήσεις λόγω οικονομίας κλίμακας διότι θα μπορούσαν για παράδειγμα να έχουν κοινέ διοικητικέ δομές και κάτι που είναι πιο πολιτικό. Μια άλλη δυνατότητα θα ήταν ότι τα τέλη αυτά για τις υπηρεσίες που κάνουν αυτές οι υπηρεσίες, αυτά τα fees, να σχεδαστούν έτσι ώστε να καλύπτουν συνολικά το κόστος λειτουργίας, όπως συμβαίνει για πολλές τέτοιες υπηρεσίες που γίνονται σε επίπεδο χωρών. Οπότε θα είχαμε και εδώ εξοικονομίες. Γιατί όχι. Γιατί όχι τα τέλη να καλύπτουν συνολικά το κόστος λειτουργίας. Αν είναι καλή υπηρεσία, αν είναι αναγκαία η υπηρεσία που είναι, γιατί αυτοί οι οποίοι ωφελούνται από αυτή την υπηρεσία να καλύπτουν όλο ή σχεδόν όλο το κόστος λειτουργίας των. Πιστεύω ότι τα θέματα αυτά πρέπει να εξεταστούν. Και συμφωνώ ότι η μελέτη αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους άλλους οργανισμούς και φορείς της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μαργάλ. Ο κύριος Ντονάνο. Θα ήθελα να μάθω γιατί επελέγησαν αυτοί οι 7 οργανισμοί. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Άλλες παρατηρήσεις. Δεν βλέπω. Ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι για το αποτέλεσμα να πω καταρχάς. Γιατί βέβαια θα ήμουν ιδιαίτερα απογοητευμένος εάν ε, το πόρισμά σας ήταν ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς ήταν πιο δαπανηροί και λιγότερο αποτελεσματικοί από τις εθνικές υπηρεσίες. Τώρα ερωτήσεις σχετικές με αυτά που είπε και ο κ. Μαραγάου. Μια άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να τεθεί είναι ποιο είναι για ορισμένους από αυτούς τους φορείς, όχι για όλους, αλλά για ορισμένους από αυτούς τους φορείς, ποιο είναι το συμπληρωματικό κόστος που προκύπτει από την ίδρυση ενός τέτοιου φορέα ενώ κάποια από τα καθήκοντά τους θα μπορούσαν να εκτελούνται από την ε, δημόσια διοίκηση. Δεν αφορά όλους τους φορείς, αλλά ορισμένους. Σχετίζεται με την ερώτηση του κυρίου Μαραγάλ. Γιατί βλέπω ότι αυτό το θέμα δεν έχει τεθεί στην έκθεση. Υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου χρειάζεται αυτόνομη αρχή που να μην ελέγχονται από τη δημόσια δίκηση, αλλά για άλλους τομείς δεν είναι αναγκαίο αυτό. Και δεύτερον, για το κόστος. Εδώ λέτε ότι για τον προπολογισμό της Ένωσης, σε σύγκριση με τα κράτη-μέλη, μειώνεται λοιπόν από το ότι υπάρχουν τέλη, ότι οι χρήστες πληρώνουν αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις υπηρεσίες. Αλλά αυτό δεν ισχύει για ορισμένου τέτοιου φορεί, οι οποίοι δεν λαμβάνουν τέτοια τέλη. Η ίδια είναι η συλλογιστική. Θα ήθελα να με πείσετε γιατί δεν είμαι μέχρι στιγμής πεισμένο. Θέλει κάνει άλλο το λόγο, όχι. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, θα μιλήσω κι εγώ θεωρείτε ότι μπορέσατε να διαπιστώσετε ότι αυτοί οι φορείς έχουν πραγματική αιτία ύπαρξης γιατί ορισμένες φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι κάθε τέτοιος φορέας κάποιοι τέτοιοι φορείς ιδρύθηκαν για να ευχαριστήσουν κάποια κράτη-μέλη έχουν συγκεκριμένη λοιπόν ε, συγκεκριμένο λόγο ύπαρξης και θεωρείτε ότι όταν υπάρχουν ε, τέτοιοι ευρωπαϊκοί φορείς αυτοί καθιστούν περιτές πλέον τις εθνικές υπηρεσίες ή τη δημόσια δίκηση γενικά ότι δηλαδή θεωρείτε ότι έτσι έχουμε εξοικονομήσεις, έχουμε και χαμηλότερο κόστος και αύξηση της αποτελεσματικότητας. Και όπως θα συμφωνούσε και ο κύριος Μαραγάλ, ένας ε, οργανισμός που τώρα λέγεται οργανισμός διανοητικής ιδιοκτησίας έχει πλεονάσματα. Και όταν είπαμε ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν πλεονάσματα, Μα είπαν όχι δεν πρέπει να γίνει αυτό γιατί αυτό θα ήταν αθέμητο ανταγωνισμός για τις ε, ε, παρόμοιες εθνικές υπηρεσίες. Συμφωνείτε με αυτή τη λογική. Κύριε Μάλαν, παρακαλώ απαντήστε σε όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Αλλά αρκετά σύντομα σας παρακαλώ γιατί έχουμε πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως ε, να επιλέξω κάποια ερωτήματα, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα που εντάξει δεν είναι τόσο σημαντικά για να απαντηθούν. Νομίζω λοιπόν ότι πράγματι είναι αλήθεια ότι ε, όσον αφορά στην απόδοση των οργανισμών αυτών, ε, κάποιοι εξ αυτών μειώνουν τον ε, προπολογισμό του και νομίζω ότι βελτιώνεται η απόδοσή του. Αλλά το τελευταίο που θα λέγαμε στη μελέτη μα είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο να μειωθεί περαιτέρω το κόστο των οργανισμών ή να βελτιωθεί περισσότερο η απόδοσή του. Επίση είναι αλήθεια ότι οι οργανισμοί αυτοί δεν είναι πολύ καλοί στο να παρουσιάσουν την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν. Προσφανώς, προφανώς και έχουν γίνει αξιολογήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές Συμφωνώ μαζί σας ότι οι οργανισμοί αυτοί δεν τα καταφέρνουν και πολύ καλά στο να αποδείξουν ότι προσφέρουν ε, υπεραξία στα κράτη-μέλη. Το ερώτημα του κατά πόσον υπάρχει ε, περιθώριο κάποιοι οργανισμοί που δεν επιβάλλουν εισφορές στα μέλη τους να το πράξουν στο μέλλον, κατά πόσον αυτό μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, ας πούμε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, ε, Αξιών και Αγορών, ένας από αυτούς που τους ερευνήσαμε, τους εξετάσαμε, πράγματι ασχολείται με το κατά πόσον μπορεί να επιβάλλει εισφορές σε μέλη τα οποία ελέγχει και ε, τα οποία αξιολογεί. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και πρέπει να τεθεί επιτάπητος, δηλαδή κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί μπορούν ε, να ε, έχουν κάποια έσοδα για να καλύπτουν τις δαπάνες τους από τις υπηρεσίες που προσφέρουν και όχι από τις επιδοτήσεις που τους χορηγεί ο ενωσιακός προϋπολογισμός. Και κάτι άλλο, σχετικά με τα έσοδα ε, για να ε, έχουν έσοδα που να τα ε, επιστρέφουν στον προπλογισμό. Αυτό σωστό είναι. Εγώ συμφωνώ. Ε, κατόπιν τούτου, παρότι είναι δύσκολο να ορίσει κανεί ποσοτικά τα ωφέλη από το να έχει αυτούς τους οργανισμούς ε, κατά πόσον αυτό είναι πιο επωφελές από το να γίνεται η δουλειά στα κράτη-μέλη. Είναι δύσκολο ποσοτικά να οριστεί. Ε, Παρ' όλα αυτά, Νομίζω ότι συμφωνήσαμε όλοι ότι οι αεροπορικές εταιρείε οι οποίες χρησιμοποιούν τους οργανισμούς συμφωνούν όλοι ε, συμφωνούν όλες οι εταιρείε ότι είναι χρήσιμοι αυτοί οι οργανισμοί και χωρίς αυτούς τους οργανισμούς ο κλάδος θα αντιμετώπιζε πολύ μεγαλύτερο κόστος. Παρότι σας είπα δεν είναι εύκολο να οριστούν όλα αυτά ποσοτικά, ε, παρόλα αυτά από τις αντιδράσεις ε, που είχαμε μέχρι τώρα έχουμε καταλήξει στο ότι ε, προσφέρουν σημαντικό έργο και από πλευράς κόστους. Κοιτάξτε, εγώ κύριε Πρόεδρε δεν έχω τίποτα να προσθέσω από αυτού. Πρόεδρος, μικρόφωνο παρακαλούμε, ο Πρόεδρος. Ναι, ευχαριστούμε. Ωραία, θα περάσουμε τώρα στην ε, δεύτερη ανακοίνωση. Σας ευχαριστούμε κύριε Μάλλον. Η επόμενη μελέτη αφορά το κόστος ε, των ε, πολιτικών, το κόστος κάθε ευρώ από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διάφορα κράτη-μέλη. Ο κύριος Μόρισον είναι αυτός ο οποίος είναι αρμόδιος ε, για την ε, ε, μελέτη αυτή και θα του δώσω του λόγο για κάποια εισαγωγικά σχόλια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα που εκπώνησε αυτή τη μελέτη για το κόστος που πληρώνουν ε, οι δικαιούχοι και οι εθνικές αρχές ε, για να υπάρχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που κάνατε εσείς ε, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη, διότι η ομάδα των ερευνητών που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό χρειάστηκε να λάβει πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να το επισημάνω εδώ. Οι γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν κάποιες επιφυλάξεις να δώσουν ε, στην ομάδα της μελέτης ε, τις ε, συγκεκριμένες πληροφορίες που χρειάζονταν προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους και χάρη στη δική σα την παρέμβαση και στη στήριξη της Αντιπροέδρου ε, Γεωργίευα καταφέραμε να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες ε, οι ερευνητέ. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο κυρία Γεωργίευα για τι προσπάθειε, της η οποία εξασφάλισε τις πληροφορίες αυτές ώστε να υλοποιηθεί μελέτη και να μπορέσουμε να επιτρέψουμε και στο Κοινοβούλιο να ε, κάνει ε, αυτό που το αναλογεί, δηλαδή τον έλεγχο της, ε, του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της μελέτης ήταν να δούμε το κόστος που πληρώνουν οι δικαιούχοι και οι εθνικές αρχές προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να προσπαθήσουμε να έχουμε και κάποιες πληροφορίες για τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των προγραμμάτων που είναι ε, στην άμεση διαχείριση και στην ε, συνδιαχείριση. Ε, αν υπάρχει πολύ ψηλό κόστος για το δικαιούχο σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίω όσον αφορά το συνολικό ποσό το οποίο θα λάμβαναν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αν το γραφειοκρατικό άρθος και το κόστος τελικά σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιους τομείς πολιτικής είναι τόσο υψηλό που δεν ενθαρρύνει τους δικαιούχους να κάνουν έτσι για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και υπήρχαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα εδώ. Για τα προγράμματα βέβαια της άμεσης διαχείρισης, όπου είναι πάρα πολύ ε, υψηλές οι κλίμακες, ε, είναι σαφές ότι το κόστος ε, για αίτηση χρηματοδότηση σε σχέση με το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι πολύ μικρότερο από το κόστος και τη συνολική κλίμακα ενός προγράμματος για μια μικρομεσαία επιχείρηση ή για κάποιο πολύ μικρή επιχείρηση. Βεβαίως η μελέτη αυτή σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται συνολική αξιολόγηση του τι γίνεται με το, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, απλώς εντοπίζει κάποια κενά και προτείνει κάποιες λύσεις ε, για την, ε, και κάποιες βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων μας και να είμαστε βέβαιοι ότι τα χρήματα φτάνουν στους δικαιούχους με πιο εύκολο και πιο γρήγορο τρόπο αλλά βέβαια όλα αυτά στα πλαίσια της υγιούς ε, ε, χρηματοπιστωτικής διαχείρισης και φυσικά ε, να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πατάξουμε την απάτη όπου υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε, θα ο περιθώριο στην παρουσίαση και θα, στη συζήτηση περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ λοιπόν από τους ερευνητές της μελέτης να μας την παρουσιάσουν και να μας πούν τα διάφορα στοιχεία. Ποιος θα πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ να σας παρουσιάσω τα βασικά πορίσματα αυτής της ε, σημαντικής ε, έρευνας κατά επόμενα 15 λεπτά. Ο στόχος της μελέτης είναι να κατανοήσουμε το κόστος το οποίο έχει σχέση με τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις και να υποβάλουμε επίσης συγκεκριμένες προτάσεις. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο και έχουμε υπολογίσει το κόστος με βάση δεδομένα τα οποία λάβαμε από τα κρατημέλη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από δικαιούχους. Με βάση όλα αυτά καταλήξαμε στο να διατυπώσουμε συγκεκριμένες συστάσεις, οι οποίες θα παρουσιάσω στο τέλος της έκτης. Επίσης θέλω να σας πω ότι η μελέτη βασίζεται σε μια επιλογή προγραμμάτων και βασίζεται στην ε, αποτελεσματικότητα ε, στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και επίσης και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Προφανώς όλα αυτά από κοινού καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα ε, του συνόλου των, της καταβολής ενισχύσεων, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ε, όπως ξέρετε λοιπόν όλοι πάρα πολύ καλά, η απλούστευση, η εναρμόνιση των ε, κανονισμών και η χορήγηση των ενισχύσεων, αυτά όλα δημιουργούν πολλές ανησυχίες στους δικαιούχους. Ήταν μια μεγάλη ανησυχία για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχουν γενικοί κανόνες, ε, συγκεκριμένοι κανόνες οι οποίες ε, διέπουν την χορήγηση των ισχύσεων. Βεβαίω και υπάρχουν σημαντικές ε, διαφορές ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα, αλλά παρόλα αυτά είναι σαφές ότι οι χρηματοπιστωτικοί κανονισμοί καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές και υποβάλλουν συστάσεις για να υπάρχει ένα υγιές περιβάλλον. Πέρα από όλα αυτά, κάθε μεμονωμένο πρόγραμμα ε, διέπεται από τους δικούς του τους κανόνες. Αυτοί λοιπόν οι κανόνες λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στοιχεία και λαμβάνουν υπόψη τους και το διοικητικό άχθος που προκύπτει. Παραδείγματο χάρη, το ότι είναι υποχρεωτικό να γίνεται αναφορά σαν παράδειγμα, νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι παράλογο το ότι ορισμένοι κανόνες διαφέρουν. Παραδείγματος χάρη είναι οι κανόνες που αφορούν την κινητικότητα για τους φοιτητές. Αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να το χειριστεί κανείς όπως ένα πρόγραμμα για ε, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ε, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει στόχος εναρμονισμού προγραμμάτων, οπουδήποτε αυτό κρίνεται κατάλληλο. Αν δούμε λιγάκι την ευρύτερη διαδικασία, θα διαπιστώσουμε ότι οι διαδικασίες μοιάζουν περίπου, παρότι όπως είπα προηγουμένως η εφαρμογή μπορεί να είναι διαφορετική. Η γενική διαδικασία και το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε βλέπετε εδώ στη διαφάνεια αποτελείται κατ' ουσίαν από τρία βασικά μέρη. Το ένα είναι η πρόσκληση ενδιαφέροντος, μετά είναι η ε, εφαρμογή και τέλος πώς κλείνει το όλο θέμα της ενίσχυσης. Ε, υπάρχει επιμερισμό διαχείρισης, υπάρχουν πολλές μορφές διαχείρισης, αλλά και ο ρόλος των εμπλεκομένων είναι διαφορετικός. Υπάρχουν γενικές διευθύνσεις, ε, ε περιφέρειες, εθνικοί οργανισμοί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε κάθε κομμάτι της διαδικασίας έχουμε τον δικαιούχο ο οποίο βεβαίω και εμπλέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Στην αρχή τη διαδικασία, σα είπα είναι πρόσκληση ενδιαφέροντο το να ε, προκύψουν ε, σε ενισχύσεις, να, στο τέλος να υπάρχουν διαπραγματεύσει για το πρόγραμμα. Και όλη αυτή η διαχείριση απαιτεί ε, πολλούς πόρους, οικονομικούς πόρους, αλλά και πόρους ανθρώπινου δυναμικού από όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους. Ας δούμε τώρα λιγάκι το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας επειδή τα οικονομικά συστήματα της Κομισιόν δεν μπόρεσαν να μας προσφέρουν τα απαραίτητα στοιχεία ε, και με τις απαραίτητες λεπτομέρειες το κόστος που σας παρουσιάζουμε ε, αφορά περισσότερο μελέτες περί και πρέπει να είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί όσον αφορά την επαγωγή των δεδομένων. Να ξέρετε ότι δεν έχουμε πάρει στοιχεία κόστους για το πρόγραμμα Erasmus, Erasmus γιατί αυτό δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη μας σε ενωσιακό επίπεδο και πάλι στο πλαίσιο της μελέτης. Σας είπα στην αρχή υπάρχουν κάποια προγράμματα εκτός του Erasmus ΣΥΝ. Η Ευρωπαϊκή Επιτή ε, χρησιμοποιεί περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ για να χορηγεί ενισχύσεις και για να ελέγχει τις αρμόδιες αρχές. Ε, κάναμε υπολογισμό των ποσοστών και αυτό σημαίνει ότι το άμεσο κόστος για την Κομισιόν είναι περίπου το 1% το 0,83% για την ακρίβεια του συνολικού κόστους και στην επιμερισμένη διαχείριση 0,1% του συνόλου. Το κόστος λοιπόν ποικίλει από 0,05% και μέχρι 0,9%. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη βεντάλια και Όσον αφορά τις περιπτώσεις που εξετάσαμε, στην επιμερισμένη διαχείριση έχουμε από 0,07% μέχρι 0,15%. Υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διαφορές που εξηγούνται και από το ότι σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και διαφορετικά στοιχεία που προκαλούν το κόστος. Αλλά κυρίως το μέγεθος της ενίσχυσης είναι καθοριστική σημασίας. Υπάρχουν βέβαια και άλλα στοιχεία που προκαλούν κόστος όπως ε, η αναφορά, η λογοδοσία, παραδείγματος χάρη, ο βαθμός του αυτοματισμού και άλλα. Αν δούμε τώρα πιο προσεκτικά το εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο, οι βασικές ε, δραστηριότητες μοιάζουν ε, με αυτές ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση διαχείριση. Εδώ το μέσο κόστος είναι 0,5% εδώ στις μελέτες περιπτώσεων που κάναμε εμείς οι έρευνες έδειξαν 3-10% ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αν δούμε το θέμα των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι, εμείς κάναμε κάποιες μελέτες περιπτώσεων και αυτοί κοστίζουν από το 1% και μέχρι και το 19%. Αυτό δηλαδή είναι ε, το μεγαλύτερο άνοιγμα της βεντάλιας. Οι δικαιούχοι ακόμα και αυτοί που ζητούν μικρά ποσά πρέπει να περάσουν μέσα από το σύνολο της διαδικασίας και το κόστος που προκύπτει από αυτούς είναι πολύ μεγαλύτερο αναλογικά από τους δικαιούχους που ε, ετούνται μικρότερα ποσά. Οι μελέτες περιπτώσεων έδειξαν ότι η διαδικασία αυτή είναι περίπου το 20 μέχρι 30% του κόστους που προκύπτει συνολικά, άρα δηλαδή ακόμα και στην περίπτωση όπου οι δικαιούχοι τελικά δεν λαμβάνουν ενισχύσεις, παρόλα αυτά ε, προκαλούν σημαντικό κόστος στην όλη διαδικασία. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η Κομισιόν έχει ήδη προβεί, έχει αναλάβει ε, πρωτοβουλίες ε, απλούστευσης, αλλά στα ερωτηματολόγια τα οποία εμείς υποβάλαμε σε διάφορους οργανισμούς διαπιστώσαμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό φορο... Ε, γραφειοκρατικό άχθος σε ενωσιακό επίπεδο υπάρχουν μη εναρμονισμένες διαδικασίες υπάρχουν ε, εκ των προτέρων αξιολογήσεις του κόστους. Δυστυχώς δεν υπάρχει εναρμόνιση, υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ψηφιοποίησης, αυτοματισμού ε, και διαφορετικό βάθος των ελέγχων που διεξάγονται. Αν πάμε σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, το διοικητικό αυτό σε μεγάλο βαθμό αφορά την ε, υποβολή αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το πρίσμα των εθνικών περιφερειακών αρχών. Αναφέρεται ότι οι κανονισμοί δεν είναι σαφείς, είναι περίπλοκοι, πολλές φορές και οι έλεγχοι που γίνονται είναι χρονοβόροι. Αν δούμε τώρα το, από την πλευρά των δικαιούχων. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να είναι γνωστό ότι η διαδικασία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη για τους μικρούς ε, οργανισμούς. Αυτοί έχουν αντιμέτωποι με πολύ περιπλοκές διαδικασίες και οι νέοι ετούντες δεν έχουν καν εμπειρία μέσα σε αυτήν τη διαδικασία. Ε, ως εκ τούτου οι νέοι ετούντες ε, ενδέχεται και να αποθαρρύνονται να υποβάλουν αιτήσει ε, για απόκτηση ενισχύσεων. Εξάλλου, για τους νεοεισερχόμενους, αποθαρρυντική είναι η όλη διαδικασία το ότι χρειάζονται πάρα πολλά συνοδευτικά έγγραφα για να υποβάλουν για τους ελέγχους. Πολλές φορές οι έλεγχοι είναι τελείως διαφορετικοί όταν διεξάγονται από εθνικές αρχές από ότι όταν διεξάγονται από κοινωτικούς ε, φορείς. Πάμε στην περίοδο 17 έως 13. Πράγματι υπήρξαν κάποιες απλουστέψεις που θα είναι χρήσιμες μέχρι το 2020. Κάποιες άλλες απλουστεύσεις προβλέπονται. Ε, υπάρχουν όμως απλουστεύσεις οι οποίες αφορούν κυρίως την επιστροφή δαπανών και διάφορες μορφές ψηφιοποίησης και αυτοματισμού. Και οι προβλεπόμενες διαδικασίες απλούστευσης αφορούν κυρίως ε, τίματα κόστους, επιστροφής κόστους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, περιορισμό υποβολής εγγράφων, τεκμηρίων και εναρμόνιση των διαδικασιών ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα σε όλα αυτά, η υπήρξαν αντιδράσεις από τους δικαιούχους που δείχνουν ότι η περαιτέρω απλούστευση και η μόχλευση είναι θέματα που ίσως θα μπορούσαν να ληφθούν περαιτέρω υπόψη. Σε πέντε τομείς. Ο πρώτος αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο και τους κανόνες, περαιτέρω εναρμόνιση μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδότησης. Αυτό μπορεί να γίνει και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. Παράδειγμα, το να υπάρχει έτσι κάποια, κάποιοι γενικοί κανόνες για την επιστροφή κόστους. Δεύτερος τομέας, ψηφιοποίηση και αυτοματισμός δραστηριοτήτων. Εκεί δεν τίθεται μόνο το θέμα το ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να αυτοματοποιούνται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο αυτοματισμός, αυτός θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια σε όλους τους δικαιούχους που ενδέχεται να αποφεληθούν από όλα αυτά. Τρίτος τομέας, βελτίωση των επιχειρηματικών ή επιχειρησιακών διαδικασιών. Εδώ ε, περιλαμβάνεται η κατάργηση ενδιάμεσων εκθέσεων. Να μην υπάρχουν διπλή έλεγχοι και σε επίπεδο κράτους μέλους και σε επίπεδο επιτροπής. Ε, να γίνεται περισσότερο ψηφιοποιημένη υποβολή εγγράφων. Τέταρτος τομέας, εξορθολογισμός ε, κάποιων διαδικασιών για την λογοδοσία και τέλος ε, μπορεί να βελτιωθεί και το σύστημα ενημέρωσης για να διευκολύνεται η όλη διαχείριση του συστήματος και για να είναι πιο εύκολο να εστιάζει κανείς την προσοχή του σε θέματα όπου μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση κόστους. Για να ολοκληρώσουμε, η έρευνά μας κατέδειξε ότι η διαδικασία χορήγηση ενισχύσεων μπορεί να πλουστευτεί περαιτέρω, θα βελτιωθεί το κόστος ε, που αφορά στην Κομισιόν, αλλά και αυτό που αφορά στα κράτη-μέλη και στις περιοχές, στις περιφέρειες, με συγχωρείτε. Πρέπει να επισημάνουμε, όλη η διαδικασία μπορεί να πλουστευτεί περαιτέρω ε, και αυτό θα ωφελήσει ε, και τους ετούντες και τους δικαιούχους. Θα περιοριστεί το γραφειοκρατικό άχθος ε, είτε εκλαμβάνεται ως τέτοιο, είτε εκλαμβάνεται ως κόστος. Και με αυτά τα λόγια επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Euh, Ευχαριστώ για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική εκθεσή σας για τις, ε, τους μεγάλους άξονες της απλούστευσης. Βεβαίως, ε, είναι σωστή η διαχείριση του προπολογισμού. Είναι τόσο περίπλοκη η διαδικασία υποβολή αιτήσεων που πολλοί εγκαταλείπουν την προσπάθεια και έτσι έχουμε οικονομίε. Αλλά έχουμε φτάσει στο όριο του παραλογισμού. Όταν πραγματικά βλέπουμε τι διαδικασίε είναι αυτέ, ελπίζω λοιπόν η μελέτη σας να βοηθήσει. Λοιπόν, ο πρώτος λόγο είναι ο κύριος Ashworth. Ευχαριστώ για την ε, πολύ χρήσιμη πληροφόρηση. Αυτό το, αυτή η διαφοροποίηση κόστους μεταξύ τομέων. Θα ήθελα μερικά περισσότερα παραδείγματα. Για παράδειγμα, από κράτος ε, μέλος στα άλλα είδατε ας πούμε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος μια περιφέρεια να είναι πιο ακριβές ή κάποιος τομέας πολιτικής υπάρχουν τομείς όπου είναι πιο μεγάλο το κόστος είναι πιο ακριβά για να υποβάλει κανείς αίτηση ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις και οπωσδήποτε αυτό μας ανησυχεί θα θέλαμε να το ξέρουμε αλλά σε άλλους τομείς θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι είναι τόσο ακριβή υποβολή αιτήσεων που είναι πολύ μικρό το... είναι πολύ μικρή η προστιθεμένη αξία. Έχετε παρατηρήσει παρακαλώ επ' αυτούν. Ευχαριστώ κύριος Μαραγάο. Με ακούτε? Τρεις ερωτήσεις. Νομίζω ότι έμεσα το είπατε κι εσείς. Προηγουμένως ε, μιλούσαμε για το κόστος των μη φορέων. Ίσως εδώ να υπάρχει κόστος ε, της έλλειψης ε, προδιαγραφών. Διαλειτουργικότητα. Πριν από λίγο το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια έκθεση για τα προγράμματα διελτουργικότητας μεταξύ λογισμικών, μεταξύ κρατών, δημοσίων διοικήσεων. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη βέβαια για να βελτιστοποιήσουμε αυτή την κατεύθυνση για τη διαχείριση των ε, επιδοτήσεων. Επιπλέον, ο κόστος του χρόνου. Δεν άκουσα να πείτε τίποτα γι' αυτό. Πόσο κοστίζει το ότι από τη στιγμή που ξεκινάει η διαδικασία μέχρι να χορηγηθεί η επιδότηση περνάει τόσος χρόνος και αναπερίπτωση πόσο, πόσος χρόνος περνάει ανα, ανα τομέα πολιτικής. Στην Ήτρε συζητούσαμε για την αναθεώρηση του ορίζοντα 2020 και άκουσα να λένε τα πανεπιστήμια και επιχειρήσεις ότι είναι ιδιαίτερα λυπηρή η κατάσταση. Έχουμε πει επανειλημμένο ότι υπάρχει γενικά θέμα νοοτροπίας των δημοσίων διοικήσεων. Η νοοτροπία τους είναι ex ante, να τα ελέγχουν όλα πριν ξεκινήσει μια διαδικασία. Ενώ η αγγλοσαξονική νοοτροπία είναι ex post, πολύ περισσότερο. Μήπως θα μπορούσαμε εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Για ορισμένα θέματα, για ορισμένους τομείς θα μπορούσαμε να μειώσουμε το κόστος και να κερδίσουμε χρόνο και να μειώσουμε την γραφειοκρατία εάν ε, εφαρμόσουμε με βεβαίως ε, προϋποθέσεις και με κοινή λογική ε, να εφαρμόσουμε λοιπόν ένα σύστημα ex post και όχι ένα σύστημα εκ των προτέρων ελέγχου των πάντων. Πρόεδρος, η κυρία Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστούμε για την μιλή, δεν την άκουσα όλοι. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, σε ε, νοσιακό επίπεδο εδώ υπάρχει ένας τεράστιος μηχανισμός όσον αφορά την επεξεργασία των αιτήσεων. Δηλαδή, ε, συγκεντρώνονται τα χρήματα για να σταλούν στα κράτη-μέλη Αυτά συνδέονται με νομοθεσία, με στόχους, με χρήση. Βεβαίως και αυτό είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία και πρέπει να είναι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Μόνο το ερώτημα που τίθεται είναι μήπως ήταν πιο σκόπιμο να λέμε ότι κοιτάξτε, Κρατήστε τα χρήματά σας, αλλά αν το πούμε αυτό, τι θα γίνει τότε με την Ένωση και το νοσιακό επίπεδο. Σας προειδοποιώ να μην ε, διατρέξουμε κίνδυνο μέσα από αυτή τη διαδικασία όπου ορίζονται κανόνες για το πώς εκταμιεύονται τα χρήματα να μην κάνουμε το λάθος να πιστεύουμε ότι μπορούμε όλα αυτά να τα πλουστεύσουμε σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τα κονδύλια για οτιδήποτε επιθυμούν. Αυτό είναι επικίνδυνο και σας το επισημαίνω. Και δεν ξέρω αν όλοι ξέρουν το τι θέλουν να κάνουν και το τι κάνουν. Δηλαδή, αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν ενισχύσεις στον προεπλογισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει αυτή η δυνατότητα τίθεται το ερώτημα μήπως ε, θα πρέπει μόνοι μας ε, να μην ε, καταλήξουμε στο να βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Γιατί ας πούμε στη Γεωργία με το πρασίνισμα τα κάναμε τόσο πολύ δύσκολα που καταλήξαμε σε κάτι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό που έπρεπε. Αν είχαμε πει Κοιτάξτε, κάντε κάτι και ε, νομίζω ότι ε, αν επικρατούσε η λογική όλοι θα ήταν ευχαριστημένοι με λίγους κανόνες, κάτι θα γινόταν. Τι θέλω να πω, ότι Πρέπει να είναι σαφές ε, τι κανόνες ορίζουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας που θέλουμε να επιτύχουμε με τις ενισχύσεις και να ξέρουμε κατά πόσο είμαστε πρόθυμοι να παραιτηθούμε από κάποιες διατάξεις. Εγώ ας πούμε είμαι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ εδώ στην αίθουσα που επίση είναι και αν υπάρχουν ε, πολλές διατάξεις πρέπει κάπως να ελέγχουμε κατά πόσο εφαρμόζονται οι διατάξεις. Αλλιώς τι να τις κάνουμε είναι θέμα συνέπειας. Γι' αυτό λοιπόν τουλάχιστον να ξέρουμε ποιο είναι το αντικείμενο της κουβέντα. Εγώ θα ήμουν ευγνώμων αν το ξέραμε. Και επίσης ε, ε, να πούμε ότι εντάξει δεν μπορούμε ε, να αφήσουμε τα πράγματα να προκύψουν όπως προκύψουν. Σίγουρα κάπως πρέπει να τα περιορίσουμε. Ας πάμε στον τομέα της έρευνας που το θίξατε. Ξέρετε, Δεκατρία δις και 7 εκατομμύρια δεν ξέρω αν το δει κανείς ποσοστιαία, κάτι γίνεται. Και στον αγροτικό τομέα είναι 5 μέχρι 7% το κόστος και δεν είναι τεράστιο το κόστος για όλο αυτό το μηχανισμό που λειτουργεί. Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσον βοηθάνε οι αριθμοί για να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς. Πάντως η μελέτη είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί η μελέτη ε, προσπαθεί όλα αυτά να τα καταστήσει κάπως χρήσιμα στο πλαίσιο του προεπολογισμού. Βεβαίως, ούτως ή Βεβαίω, ούτω ή άλλω ζούμε στην πραγματικότητα. Είναι πολύ επίκαιρο αυτό. Είστε εισηγήτρια εξ ονόματο Επιτροπή ε, Προπολογισμών του Omnibus ε, για την απλούστευση του δημοσιονομικού κανονισμού. Επομένω, η μελέτη αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει. Ο κύριο Ντονανό. Ακριβώς οι διαδικασίες είναι αυτές οι οποίες συζητούμε. Αν έχουμε 27 δις ε, διαρθρωτικών τομείων που δεν χρησιμοποιούνται γιατί δεν υπάρχει υλοποίηση, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Επειδή εγώ ε, γνωρίζω τα πράγματα εδώ και χρόνια, ξέρω πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα δεν ξεκινούν γιατί οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ ε, σύνθετες. να ελέγχουμε εκ των υστέρων, εκ των προτέρων, κατά τη διάρκεια, αλλά δεν θα λειτουργήσει έτσι η Ευρώπη. Και νομίζω ότι σήμερα, λαμβάνοντα υπόψη και αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, δεν χρειαζόμαστε τέτοια πράγματα. Πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε να έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι πρέπει να μπορούμε να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία θα δίνουν τις μεγάλες κατευθύνσεις και τα ευρωπαϊκά ε, στοιχεία και από εκεί και πέρα να κάνουν τα κράτη αυτό που τους αναλογεί χωρίς να γίνεται συνεχής έλεγχος, απλώς ένας έλεγχος εκ των υστέρων στο τέλος, στο σημείο της παράδοσης. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα θέμα εγώ κρυώνω γιατί νιώθω σαν να είμαστε σε ένα ψυγείο. Δεν έχει μόνος εδώ. Θα και ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω αν κάνουμε οικονομία στη θέρμανση εδώ. Ναι, πάντων, αν κάνουμε, τουλάχιστον κάνουμε αποταμίευση. Λοιπόν, το θέμα είναι ζωτική σημασία. Είναι τόσο σύνθετο που ορισμένε φορέ πρέπει να ζητήσουμε μελέτη για να μπορέσουμε να κατατηρήσουμε τα σφακέλου με τα θέματά μα. Τι κάνετε εσεί. Ε, ε, φαντάζομαι ότι και εσείς ε, ανατρέχετε σε κάποιους πότε πότε ουσιαστικά καταστρέφεται ένα τμήμα της αγοράς ε, του γραφείου σας. Και εδώ ε, απαντώ σε συνέχεια των όσων είπε η κυρία Γκρέσλε, αλλά θα πρέπει να ξαναδούμε τους κανόνες. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα είναι κάτι πειραματικό, καινοτόμο και τελικά φτάνουμε σε ένα σημείο που τα ε, ισοπεδώνει όλα και δεν γίνεται τίποτα. Είναι πολύ αποτελεσματικό αυτό γιατί αποταμιεύουμε πολλά χρήματα, αλλά δίνεται μια εικόνα ε, τελείως καρικατούρας της Ευρώπης και υπάρχει απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης. Μήπως μπορούμε λοιπόν να τα διαβαθμίσουμε κάπως για κάποια προγράμματα, να ε, ελαφρύνουμε λίγο την χαρτούρα και τη γραφειοκρατία. Ε, φαίνεται ότι ορισμένες φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να καθυστερήσει τα πάντα και είμαστε στα όρια της καρικατούρας και δίνουμε μια πραγματικά επωνύδιστη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού μπορούμε να φτάσουμε λοιπόν προκειμένου να πλουστεύσουμε τα πράγματα, λαμβάνοντα υπόψη βέβαια και το εθνικό επίπεδο και το τοπικό επίπεδο, γιατί εγώ επισκέφθηκα κάποιε περιοχέ στη Γαλλία παραδείγματο χάρη στην περιοχή του Λίγυρα ε, και επισκέφθηκα οι ε, υπηρεσίε που ήταν αρμόδιε για ε, τέτοια πράγματα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και πραγματικά δημιουργούν την απασχόληση, αλλά πραγματικά η γραφειοκρατία είναι τόσο πολύ που δίνει μια πολύ ζωφερή εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη, για πιστώσει για το Εράσμου θα μπορούσαν ίσω να υπάρχουν πιο απλές διαδικασίες. Ε, συνέχεια προσκλήσει υποβολή προφορών ε, με πολύ μεγάλους περιορισμούς. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου πραγματικά ε, θα πρέπει να σταματήσουν τα προγράμματα. Δεν μπορούμε να δώσουμε λίγα χρήματα. Πρέπει να υπάρχει μια κλιμακωτή διαδικασία. Δεν μπορούμε να ζητούμε τεράστιο αριθμό χαρτιών για να πάρει κάποιο χρηματοδότηση για αδελφοποίηση των δήμων μεταξύ δύο διαφορετικών χωρών, ε, οι ε, τοπικές αρχές θα πούνε ότι εντάξει το είδαμε, πήρανε βαθμό 50 στα 50, στα 100, αλλά για να πάρουν ε, χρηματοδότηση πρέπει να έχουν 75 στα 100 παραδείγματος χάρη. Αυτό τους αποθαρρύνει και στη συνέχεια δεν κάνουν αιτήσει. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τι θα έχουμε στα χέρια μας για να εξετάσουμε το όμνιμπους που θα έρθει. Όλοι αυτοί εκ των προτέρων έλεγχοι για παράδειγμα. Ξέρω ότι ορισμένε φορές δεν προχωρούμε γιατί σταματάνε αμέσω. Ε, όλοι αυτοί οι οποίοι θα ε, μπορούσαν να είναι ε, αυτοί οι οποίοι θα έδιναν κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ζέμα. Η κυρία Γκρέσλε. Just Μία παρατήρηση. Κατά τη γνώμη μου, ακόμη και το πιο ακόμη και για το πιο μικρό πρόγραμμα όσο πιο μικρό είναι το πρόγραμμα τόσο πιο μεγάλο είναι το διοικητικό κόστος εάν για το ΣΕΦ το κόστος είναι 0,0005 τότε δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά έχουμε τόσο πολλά προγράμματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Άρα καλύτερα θα ήταν να μην έχουμε μικρά προγράμματα, αλλά μέσω μικρών προγραμμάτων πλησιάζουμε τους πολίτες. Αν ο στόχος μας είναι να έχουμε μόνο μεγάλης διάστασης προγράμματα, θα έπρεπε να εκπαιδεύσουμε και τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις, αλλά οι κανόνες μας δεν είναι ε, σταθεροί. Κάθε πέντε χρόνια ε, θεωρούμε ότι είναι η ιερή υποχρέωσή μας να αλλάζουμε όλους τους κανόνες. Αντίθετα, θα έπρεπε να υπάρχει σταθερότητα των κανόνων για να συμβάλλουμε σε καλύτερη Ευρώπη και να διορθώνουμε μόνο ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο. Αλλά εμεί κάθε πέντε χρόνια τα αλλάζουμε όλα. Γιατί σε κανένα κράτος μέλος δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα των κανόνων. Έτσι θα μπορούσαν και οι εθνικές διοικήσεις να μαθαίνουν να τους εφαρμόζουν. Το χειρότερο από τα προγράμματα που έχω παρακολουθήσει είναι το Leader που γίνεται για μικρέ ενώσεις, φορεί και εκεί λέμε και ε, τελικά δεν φτάνουμε σε αυτές τις μικρές οργανώσεις γιατί είναι τόσο περίπλοκες οι διαδικασίες. Οι οργανώσεις αυτές τις μικρές μια φορά στη ζωή τους θα κάνουν τέτοια αίτηση. Δεν έχει έννοια λοιπόν. Πρέπει νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο ταπεινόφρονες για τον τρόπο με τον οποίο να αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Έτσι θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αλλά θεωρούμε ότι η εθνική διοίκηση επίσης δεν ξέρει πώς να διχειριστεί τα προγράμματα. Δεν υπάρχει ηγεσία. Δεν υπάρχει κάποιος που να αναλαμβάνει πρωτοβουλία και να δίνει εντολές. Ή κάθε 5-7 χρόνια. Και τελικά αυτή είναι η δουλειά μας, να αλλάζουμε τους κανόνες. Αυτό ισχύει και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά είναι στα όρια της γεωγραφίας, της καρικατούρας έχουμε την εντύπωση ότι ακόμη και το πιο ανόητο πρόγραμμα, εάν έχει εφαρμόσει ε, τυπικά τους κανόνες, ε, θεωρείται θαυμάσιο. Και μπορώ να σας δώσω παραδείγματα από προγράμματα που έχω ελέγξει επί τόπου. Ωραία. Ε, μπορείτε να μας πείτε και εσείς ποια είναι, ποια είναι η αντίδρασή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κάποια σχόλια, ξεκινώντας από τις τελευταίες ε, ερωτήσεις. Είπατε ότι πρέπει να απλουστευτεί η διαδικασία. Νομίζω ότι όπως λένε και τα πορίσματα της μελέτης μας, υπάρχει περιθώριο, σημαντικό περιθώριο βελτίωσης και πολλές από αυτές τις ενδεχόμενες απλουστεύσεις εγκρίνονται από όλους τους εμπλεκόμενους με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Υπάρχει ότι συμφωνία μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Εάν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν αυτές τις διαδικασίες εντελώς, να είναι πολύ απλούστερη διαδικασία, αλλά επ' αυτού, ε, εάν θέλετε να έχετε μια διαδικασία διαχείρισης επιδοτήσεων, ε, πρέπει να την έχετε. Είναι η καλύτερη αυτή που υπάρχει τώρα. Δύσκολο να το κρίνει κανείς, όπως είπα. Είναι πολύ διαφορετικέ οι διαδικασίε ανάλογα με τα προγράμματα, βασίζονται σε διαφορετικού κανόνε, διαφορετικού κανονισμού, Άρα με τι να τα συγκρίνεις στον υπόλοιπο κόσμο για να πει ποιε είναι τιμέ αναφορά να βαθμολογήσετε την απόδοσή σα. Έχουμε την καλύτερη δυνατή διαδικασία. Σίγουρα όχι. Υπάρχει περιθώριο βελτίωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ισχύουσα δεν έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσει ανάλογα με τις προσδοκίες. Για ένα άλλο σχόλιο, εάν οι δικαιούχοι φέρουν τμήμα του κόστους, ναι, έχουν κάποιο κόστος, έχουν το προσωπικό τους που ασχολείται με αυτή τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος και συχνά λαμβάνουν και τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων γιατί είναι περίπλοκη διαδικασία. Αυτό σημαίνει τότε ότι πραγματικά πληρώνουν επιπλέον Κόστο σε κάποιον άλλον, όλα αυτά συνυπολογίζονται στα ποσοστά κόστο που αναφέραμε. Υπήρξε ένα σχόλιο, μήπω είναι υπερβολικά εξάντε η προσέγγιση μας από την πλευρά των δικαιούχων, θεωρούν ότι εξάντε πρέπει να υποβάλουν πολύ αναλυτικούς φακέλους και θεωρούν ότι κατόπιν επίσης γίνονται πολλοί έλεγχοι. Ακόμη και χρόνια μετά την ολοκλήρωση του προγράμματός τους χρειάζεται για παράδειγμα να υποβάλουν κάποια δικαιολογητικά, γίνεται ένα συμπληρωματικό έλεγχος για να μην αναγκαστούν να επιστρέψουν ένα τμήμα τη επιδότηση. Είναι λοιπόν και στην αρχή και στο τέλος βαριά η διαδικασία. Για τις προηγούμενες τώρα ερωτήσεις για το εάν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορέ του επίπεδου κόστου από χώρα σε χώρα, δεν μπορέσαμε να συλλέξουμε επαρκή στοιχεία από όλα τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή σύγκριση αλλά εξετάζοντας έτσι δειγματοληπτικά τα στοιχεία που λάβαμε για τα διάφορα προγράμματα τότε νομίζω ότι αυτό που ανέφερε ο συνάδελφός σας ισχύει. Για παράδειγμα η διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη έχει μέσο επίπεδο επιδότησης 37 εκατομμύρια και εδώ υπολογίσαμε ότι το κόστος είναι 0,05 αναλογικά, πρόεδρος, διακόπτη, να σας διακόψω. Ορισμένοι από αυτούς τους συμβούλους ε, λαμβάνουν μία επιπλέον αμοιβή εάν ε, εγκριθεί ε, η επιδότηση. Ξέρετε ποιο είναι το ύψος. Απάντηση όχι. Δεν έχουμε καμία... Ε, δεν έχουμε στοιχεία για το τι, ποιος, ποιο είναι το ύψος αυτής της ε, αμοιβή έγκρισης. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε λοιπόν. Δεν ήταν τμήμα της μελέτης μας. Για να συνεχίσω για την ερώτησή σας. Διαπιστώνουμε λοιπόν υψηλού βαθμού συσχέτιση μεταξύ του επίπεδου της επιδότησης και του ποσοστού κόστους. Άλλο παράδειγμα. Το πρόγραμμα ΕΑΣΥ όπου το κόστος είναι υψηλό, 9,6% της επιδότησης. Εδώ όμως ε, το μέσο επίπεδο επιδότησης είναι 400.000. Ορίζον 2020, μέση επιδότηση 1,7 εκατομμύρια. Το κόστος είναι κάπου ανάμεσα. Είναι περίπου 2%. Αν το εξετάσω λοιπόν από την ε, οπτική γωνία του δικαιούχου, γιατί εξετάσαμε επιδοτήσεις διαφόρων ε, επιπέδων, για τον ορίζοντα 2020 είχαμε πει για μια συγκεκριμένη περίπτωση ε, είχαμε μια επιδότηση 1,5 εκατομμύριο και το κόστος ήταν περίπου 10%. Μια άλλη επιδότηση 60.000 ευρώ, πολύ μικρή επιδότηση, του EASF του ESF, του, Κοινωνικού Ταμείου. Και εδώ το κόστος για το δικαιούχο ήταν 20%. Πολύ σημαντική λοιπόν η σχέση μεταξύ του ύψους της επιδότησης και του κόστους. Από την οπτική γωνία λοιπόν του δικαιούχου και επειδή δεν εγκρίνονται όλες οι επιδοτήσεις για ορισμένα προγράμματα μόνο το 10% ενώ για άλλα το 90% των αιτήσεων εγκρίνονται Εάν λοιπόν συνυπολογίσουμε το κόστος για όλων, για όλους τους ετούντες που δεν λαμβάνουν τελικά επιδότηση, συνολικά το κόστος για όλους τους ετούντες κατά μέσο όρο είναι ε, πολύ υψηλό. Μα είναι άπειρο λέει ο πρόεδρος. Όταν έχεις δαπανίσει ένα ποσό και δεν παίρνεις τίποτα, είναι άπειρο. Ολοκληρώσατε. Με βάση τις περιπτώσεις που εξετάσαμε, είπαμε ότι είναι μεταξύ 20 και 30%. Εμείς βέβαια οι περιπτώσεις που εξετάσαμε ήταν όλες επιτυχείς αιτήσει. Αλλά είπαμε ότι συνολικά το 20-30% της δαπάνης που πρέπει να κάνουν είναι κόστος υποβολής της αίτησης. Είναι λοιπόν γύρω στο 20 με 30% του κόστους Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Πρέπει κάπως να το ε, διαβιβάσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι κάνουμε έργο προπολογισμού, κυρία Γκρέσλε. Η έλεγχη που θα κάνουμε εκ των υστέρων, να κατάλαβα καλά. Μήπως μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση. Λοιπόν, αυτό ήταν για το κόστος εκ των υστέρων στην ουσία. Εκ των προτέρων, συγγνώμη. Αλλά από εκεί και πέρα θα γίνει και ένας έλεγχος των λογαριασμών. Εγώ ήμουν πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου και μου είπαν ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και είπα εξαιρετικό ε, και αμέσως αρχίσαμε να σκεφτόμαστε και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είχαμε 50% συγχρηματοδότηση, προσλάβαμε και ένα συνεργάτη γιατί χρειαζόμασταν εμπειρογνωμοσύνη και τελικά έπρεπε να γίνουν ε, πάρα πολλοί δαπανηροί έλεγχοι και πρέπει αυτά να τα δούμε ε, εις βάθος. Κύριε Γκρέσλε. Θα ήθελα να σας επισημάνω το εξής. Κάθε ταμείο είναι διαφορετικό. Καθένα έχει τις δικές του δυσκολίες. Δηλαδή, πριν από 10 χρόνια, μπορεί να φαίνεται παλιά, αλλά πριν από 10 χρόνια ασχοληθήκαμε με την έρευνα. Με την έρευνα και ενισχύσει για την έρευνα. Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στου κανόνε συμμετοχή. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Τώρα μιλάμε για 90 ημέρε για τη χορήγηση ε, επιδοτήσεων και αυτό σημαίνει βελτίωση. Και εγώ το 2005 είχα καταρτήσει στατιστικά δεδομένα εκεί χρειαζόμασταν 340 ημέρες, δηλαδή μέχρι και δύο χρόνια για τη χορήγηση ενισχύσεων. Άρα χάρηκα πάρα πολύ, βελτιώθηκε η κατάσταση και δεν είναι αλήθεια ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Ε, βεβαίως υπάρχει κι άλλο περιθώριο για περισσότερη βελτίωση. Πάντως μην ξεχνάτε ότι εδώ μιλάμε για λεφτά φορολογούμενου, τα οποία εκταμιεύουμε. Και τίθεται το εξή ερώτημα. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα για μένα. Αυτό που με τρομάζει, εκτός από το leader, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο γιατί εκεί πρόκειται για μικρά ποσά. Και εγώ και στη δική μου εκλογική περιφέρεια έχω κάνει μία έρευνα για τις δαπάνες έρευνα για τις ε, δαπάνες που προκύπτουν για τις τοπικές αρχές και έφτασα μέχρι και σε διοικητικό κόστος 40%. Άρα δηλαδή το 20% το θεωρώ βελτίωση. Και μπορεί να υπάρξει και πέρα ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Στο κοινωνικό ε, ταμείο πρέπει να δούμε πού ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Γιατί όλα αυτά διαδραματίζονται σε τοπικό επίπεδο Κατά τη δική μου άποψη οι συσχετισμοί είναι τελείως διαφορετικοί. Αν θέλετε επ' αυτού να συζητήσουμε, δυστυχώς οι συντονιστές δεν μου είπαν τίποτα, δεν με ενημέρωσαν επ' αυτού, αλλά και πάλι θέλω να σας πω ότι υπάρχει ο κανονισμός για τους διάφορους ε, τομείς. Λυπάμαι που πρέπει να το πω. Αυτό δεν είναι η ε, δημοσιονομική ο δημοσιονομικός κανονισμός. Στο δημοσιονομικό κανονισμό έχουμε βελτιώσεις. Αυτοί δεν πέρασαν στο κανονισμό των τομέων και γι' αυτό προέκυψε το Omnibus για να συνδεθούν αυτά τα δύο. Ε, θέλω να σας παρακαλέσω να το πείτε αυτό όταν μιλάτε για περιγραφή κόστους να μας πείτε για ποιο σύνολο ποσού μιλάτε στην περίπτωση της ενίσχυσης. Για μας είναι σημαντικό αυτό για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για το διοικητικό κόστος που προκύπτει σε σχέση με, τα, με τις ενισχύσεις. Ε, εμένα θα με ενδιέφερε να γνωρίζω αυτό το κόστος. Κατά τα άλλα, η περίπτωση αυτή που αναφέρεται σχετικά με το Περιφερειακό Ταμείο του Βελγίου ότι χρειάστηκαν 3,5 χρόνια επ' αυτού πρέπει να σας γιατί, να ρωτήσω γιατί έγινε αυτό. Ε, και αυτό είναι συνηθισμένο μάλλον διότι οι διοικήσει ε, και ε, δεν προχωράνε υπηρεσίες με τους κανονισμούς. Κοιτάξτε, ναι, αλλά είναι ουσιώδη το θέμα. Δεν θα το λύσουμε σήμερα όμω. Το Ταμείο συνοχή είναι ένα μέσο ώστε τα κράτη-μέλη να πάρουν αυτό που του αναλογεί. Τελικά δεν έχει και τόσο σημασία. Πρέπει κάπω να επιστραφούν τα χρήματα. Και υπάρχουν δύο τρόποι να ξανάρθει. Η γεωργική πολιτική και η ταμείο συνοχή. Νομίζω ότι ε, βάλαμε πλέον ε, το πόδι μας σε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θα επανέλθουμε σήμερα, αλλά κυρία Γκρέσλε με την Επιτροπή σας ίσως θα πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη δουλειά επί του θέματος. Ε, εσείς ε, κύριοι, εάν βέβαια είναι στα πλαίσια της εντολής σας, ε, θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να σας εμπλέξουμε, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες συστάσεις που διατυπώνεται. Σήμερα δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Δεν ξέρω, ο κύριο Μόρες, αν δεν ξέρω να συμφωνεί, να ε, μην τα αφήσουμε αυτό το θέμα έτσι. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Ιδίω όταν κοιτούσαμε τα θέματα ε, συνδιαχείρισης, ε, και με την ομάδα μελέτης ήταν σαφές το μοντέλο που διαπιστώσαμε. Όσο πιο μικρά ήταν τα προγράμματα, τόσο μεγαλύτερο ήταν το μερίδιο του κόστους. Και το τμήμα της λύσης θα μπορούσε φυσικά να είναι ε, να απαιτούνται κάποια διοικητικά έγγραφα ε, ανεξάρτητα από το μέγεθο τη εταιρεία. Είναι οι ίδιε οι απαιτήσει ανεξάρτητα από τι διαστάσει του προγράμματο. Ορισμένε φορέ, αν πρόκειται για ένα μικρό πρόγραμμα, αν πρόκειται ας πούμε για ένα νέο επιχειρηματία, αν όλοι οι νέοι επιχειρηματίε πρέπει να τηρήσουν τι ίδιε υποχρεώσει με πολύ μεγάλε επιχειρήσει, οι οποίε κάνουν έτσι για πολύ μεγάλα προγράμματα στο Connecting Europe Facility, ε, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Δεν μπορούν καν να κάνουν την αίτηση, αλλά μπορεί να αποτύχει και μια μικρή επιχείρηση ε, ολοσχερός. Επομένως θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με το διοικητικό άχθος, τι μπορούμε να μειώσουμε και όσον αφορά την ε, διαχείριση και τον έλεγχο, ε, συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική ε, διαχείριση για όλους τους οργανισμούς και αυτό μπορεί να γίνει μέσω κατάρτισης, κατευθυντήριων γραμμών, υλικού για το προσωπικό, για την διαχείριση των διαδικασιών επιδοτήσεων και όσον αφορά την υλοποίηση από εκεί και πέρα, να υπάρχει μια εναρμανισμένη προσέγγιση και κανόνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο, κύριε Πρόεδρε,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 ζητά συνεχώ το Κοινοβούλιο εναρμόνιση των διαδικασιών σε όλα αυτά τα προγράμματα και τι διαδικασίε χρηματοδότηση Και ήταν σωστή η εμπνευσή μα. Και φυσικά είναι σωστό που είπε και η κυρία ε, Γκρέσλε, το να είναι προβλέψιμοι οι κανόνε. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε κανόνε κάθε πέντε χρόνια. Ε, σίγουρα επιβάλλει παραπάνω ε, άχθος αυτό. Ε, και εμεί, έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά να κάνουμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και αυτή η μελέτη αποτελεί απλώ την αφετηρία τη διαδικασία. Δεν θα πρέπει αυτό το θέμα ε, να το ξεχάσουμε, να ξεχάσουμε τη μελέτη. Ε, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδύλιων. Πολύ καλά. Ολοκληρώνουμε λοιπόν έτσι. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση. Ε, Ιουνίου από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο δημοσιονομικό κανονισμό. Ε, υπάρχει και το κείμενο που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα και θα μας υποβληθεί για να το συζητήσουμε και να ψηφίσουμε μέχρι τις 30 Ιουνίου. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές διαδικασίες ε, που θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε, τις οποίες μπορούμε να ε, προτείνουμε βάσει και των συστάσεών σας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την εμπειρογνωμοσύνη σας, για τις διευκρινήσεις σας και ε, για την διάβια με την οποία μας τα παρουσιάσατε και ελπίζω να επιδείξουμε και το θάρρος να περάσουμε στην πράξη. Περνάμε τώρα στην γνωμοδότηση της κυρίας Μούντι για το η Δημιουργική Ευρώπη. Thank you very much. Uh, yes, so... Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια γνωμοδότηση λοιπόν για την Επιτροπή Πολιτισμού για το δημιουργικό κλάδο που είναι γύρω στο 4,4% του ΑΕΠ της Ένωσης. Στην γνωμοδότηση αυτή αναγνωρίζεται η απλούστευση με βάση προηγούμενες εκθέσεις μετά την ε, εφαρμογή, έναρξη εφαρμογής του το 2014 αλλά υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης στις πιστώσεις, επιτυχούς αίτησης για την απόκτηση πιστώσεων, ιδιαίτερα για πολύ μικρούς ε, φορείς ενώσεις του πολιτιστικού κλάδου στον τομέα του πολιτισμού. Βλέπω δεν υπάρχει κανείς που να έχει μείνει εδώ στην αίθουσα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η νέα δυνατότητα, η διευκόλυνση χρηματοδοτικής εγγύησης, χρηματοπιστωτικής εγγύησης, συγγνώμη. Αυτό ελπίζουμε να προσθέσει προστιθέμενη αξία και να δημιουργήσει απασχόληση, απασχόληση στον τομέα. Τα ποσοστά εκτέλεσης του προγράμματος είναι πολύ ψηλά. Αυτό σαφώς καταδεικνύει τη σημασία των εργασιών που στηρίζει και άρα την ανάγκη ύπαρξης και διατήρησης και ίσως και αύξησης της χρηματοδότησής του. Και τέλος, υπάρχει μια διαπολιτιστική διάσταση. Αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο τώρα, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, κινήσεις πληθυσμών, ιδιαίτερα με την κρίση του προσφυγικού. Πρέπει αυτό να αναγνωριστεί και να στηριχθεί ως συνιστόσα του προγράμματος. Λοιπόν αυτά και αν έχετε τροπολογίες ε, για να ολοκληρώσουμε τη γνωμοδότησή μας, για να τη στείλουμε στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μούντι. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω εδώ το κείμενό σας. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ε, ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Μαραγάλ. Όχι, όχι, θα συνεργαστώ. Θα συνεργαστώ με την κυρία Μούντι με πολύ καλή διάθεση. Διότι συμφωνούμε. Βεβαίως θα σας βοηθήσουμε. Μα όλοι νομίζω συμφωνούμε, λέει ο πρόεδρος, με την κυρία Μουντή. Λοιπόν, και ήσασταν τόσο πιστική, κυρία μου. Όλοι όσοι εκφράστηκαν και όσοι δεν εκφράστηκαν και όσοι επίσης ε, δεν παρευρίσκονται θεωρώ ότι συμφωνούν. Όλοι θέλουν να σας στηρίξουν. Χαιρετίζω το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα σύντομη και περιεκτική η γνωμοδότησή σας. Αν υπάρξουν τροπολογίες να υποβληθούν μέχρι τις 3 ώρα στις 14 ενδεκάτου για να ψηφίσουμε στις 8 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή μας η Επιτροπή Πολιτισμού, ε, υπεύθυνη επί της ουσίας, θα εκφραστεί στις 24 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Οπότε τώρα να ακούσουμε την Επιτροπή. Που θα έπρεπε να μας μιλήσει από τις 5 και 4. Και βεβαίως είναι 17 και 14. Για το πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη εκτός της Ένωσης. Θα μιλήσει ο κύριος Σιλβάνο Πρέζα που είναι αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Μπούτζα ο κύριος ε, Ριντόλφη Διευθυντή τη ε, Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ και εκπρόσωποι των άλλων γενικών διευθύνσεων που μπορεί επίση να πάρουν το λόγο είναι ο κύριο Πάλο Μάρτινς που είναι υπεύθυνο ομάδας στην Γενική Διεύθυνση ΝΙΑΡ. Λοιπόν, παρακαλώ καθίστε συνάδελφοι. Και ξέρω ότι όσοι δεν παρευρίσκονται μας παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου. Οπότε κύριε Πρέζα είστε ο πρώτος προς τον οποίο είναι στραμμένες οι κάμερες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας κάνω εισαγωγή στο σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης και θα σταθώ κυρίως στις πτυχές του προπολογισμού και θα συνεχίσω από εδώ και πέρα στα αγγλικά για να κάνω την παρουσία μου. Σύμου. Στα μέσα του Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη μέτρων για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και σε αυτή τη δέσμη μέτρων είχαμε αυτό που λέμε στην ορολογία του προπολογισμού κάποια top-up για την περίοδο μέχρι το 2020 και στον τίτλο 4 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κάποιες προσαρμογές της τάξης του 1,4 δισεκατομμυρίου ε, σε ε, δαπάνες. 220 ε, εκατομμύρια εξ αυτών είναι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα για τη δημιουργία ενός Ταμείου Εγγύησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δημιώσιας Βιώσιμης Ανάπτυξης. 115 εκατομμύρια είναι για το Ταμείο Εγγύσεων για την επέκταση του ε, κονδυλίου δανειοδότησης Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι προτάσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή και είναι υποσυζήτηση στην Επιτροπή σας αφορούν την εφαρμογή του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Σχεδίου Επενδύσεων που περιλαμβάνει την επέκταση το, εις δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και την, το ανάκτηση στο ποσό του κανονισμού για το εξωτερικό ταμείο Η Οι συνάδελφοι θα σας ε, πούν για την χρηματοδότηση των μέσων που συζητούμε στη συνέχεια. Να σας πω απλώς, πολύ σύντομα, ε, τι σημαίνει αυτό για τον προϋπολογισμό. Όσον αφορά τις δαπάνες, ο πρώτος πυλώνας ε, του Ευρωπαϊκού ε, Ταμείου Εξωτερικών Επενδύσεων είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Θα δοθούν 3,3 δις που με τη σειρά τους μέσω των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται θα οδηγήσουν σε 44 δις επενδύσεων και πολύ περισσότερα εάν υπήρχε αντίστοιχη συνεισφορά στο Ταμείο Εγγυήσεων από τα κράτη-μέλη. Από αυτά τα 3,3 δις, τα οποία ζητήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα 2 δις θα προκύψουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και τα υπόλοιπα θα δοθούν από τα προγράμματα DCAI και ENI του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Όσον αφορά τον προγραμματισμό, στην διορθωτική επαστολή παριθμών 1 στον προπολογισμό του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 250 εκατομμύρια μέσω της κινητοποίησης του αποθεματικού για το Ταμείο Εγγυήσεων και ε, μαζί με αυτό να μεταφέρουμε και 25 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας. Συνολικά, για το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονία συνολικά θα έχουμε 100 εκατομμύρια και προβλέπεται μια δόση 25 εκατομμυρίων το χρόνο για το ε, Ταμείο Εγγύησεων. Γι' αυτό στη διορθωτική επιστολή παριθμών 1 οι συνέπειε για τον προπολογισμό για αυτή τη νέα γραμμή προπολογισμού προβλέπουν την αύξηση κατά 275 εκατομμύρια. Τα 250 είναι από την κινητοποίηση του αποθεματικού και τα υπόλοιπα 25 εκατομμύρια είναι από το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονία. Οι συνάδελφοι, όπως σας είπα, θα σας πούνε τα ουσία. Η χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλειών είναι ένας συνδυασμός νέων κονδυλίων, τα οποία προέρχονται από την ευελιξία που επιτρέπεται βάσει ε, του ε, παρόντος πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, το να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο αποθεματικό όταν είναι διαθέσιμο και τη χρήση καινοτόμων μέσων, όπως για παράδειγμα την εγγύηση του ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιώσιμης ανάπτυξη. Και επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΗΝ, ε, τον κύριο Αζέν, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα βασικά ε, στοιχεία της επέκτασης αυτής της, ε, του Ταμείου Εγγύησεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το δεύτερο μέσο, έτσι. Για το πρώτο τι ε, ποσοστό έχουμε. Είπατε ότι έχουμε δύο δις από το Ταμείο Ανάπτυξης. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα. Είναι ξεχωριστό αυτός ο προπολογισμό και τον διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένω, δεν έχει κάτι να πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μα απογοητεύει αυτό. Ένα δι θα έρθει από το ε, ε, Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονέα και το DCI, το Αναπτυξιακό. Ναι, στην ε, παρουσίαση που θα σας κάνει ο συνάδελφος εντός ολίγου, θα σας παρουσιάσει τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης για αυτό το νέο Ταμείο για την ε, Βιώσιμη Ανάπτυξη και αν θέλετε βεβαίως, δεν ξέρω, μπορούμε να τα κάνουμε και τώρα. Όχι, εντάξει, μας παρουσιάσατε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης ε, και παίρνετε ένα ποσό όπως και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υπάρχει και μόχλευση, όπως και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα είναι 3,3 δις, είπαμε, και θα μας δώσουν 44 δις επενδύσεων. Θα είναι μικρότερο δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο κύριος Ζανζέλ τώρα έχετε το λόγο. Εκφίνα. Euh, ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θα σας παρουσιάσω την πρωτοβουλία για το Εξωτερικό Ταμείο και την αναθεώρηση του Ταμείου που αφορά την μακροοικονομική βοήθεια και τα εξωτερικά στοιχεία. Θα τα πω αγγλικά. Όσον αφορά τώρα ε, την εντολή ε, σχετικά με το 2004-2020, καλύπτονται εγγύησης. Ε, έχουμε μία συνολική εγγύηση που καλύπτει τα πάντα για τη δανειδότηση του ιδιωτικού τομέα. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε μόνο τον πολιτικό κίνδυνο και όχι ε, άλλε μορφή κίνδυνο. Ποιο είναι λοιπόν το βασικό στοιχείο τη ε, πρόταση, τη οποία θα σα παρουσιάσω. Έχουμε ένα νέο οριζόντιο στόχο για τη μετανάστευση, αύξηση της εγγύησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από αυτό που είχε αρχικά προβλεφτεί, ε, προβλέπουμε την περιφερειακή κατανομή και προβλέπουμε και κάποιες άλλες αλλαγές ε, που έχουν σχέση με την ευελιξία και με τις επιλέξιμες χώρες. Όσον αφορά τους ε, νέους στόχους ε, για τη μετανάστευση, έχουμε μια βασική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι η πρωτοβουλία Resilience Initiative, όπως αναφέρεται. Στόχος είναι επιπρόσθετη χρηματοδότηση για να επέλθουν ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές ποσοτικέ αλλαγέ. Εκεί προστείνουμε να, αυξηθούν, ε, να αυξηθεί το ποσό με άλλα 2 δι ευρώ να προσθεθούν άλλα 2,3 δις ευρώ, έτσι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει δραστηριότητε του ιδιωτικού τομέα προ όφελο ε, των μεταναστών και της ε, φιλοξενούσα χώρα. Πέρα από αυτά τα οποία έχουν ήδη εκταμιευτεί. Δεύτερον, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, εισάγουμε και μια ε, ποιοτική καινοτομία που προβλέπει την άμεση χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή ε, χορηγεί μια σφαιρική εγγύηση που καλύπτει τα πάντα και όχι μόνο τον πολιτικό κίνδυνο. Κάτι που μέχρι τώρα δεν το κάναμε στο πλαίσιο αυτού του μέσου. Αν δούμε λιγάκι τα στοιχεία, είναι 27 δις ε, το ανώτατο όριο του ELM, άλλα 3 δις ε, που προστίθενται για δραστηριότητες του δημόσιου τομέα προς όφελος των μεταναστών και άλλα 2,3 δις με τη μορφή εγγύησεων που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα ως ένα τμήμα του τήρητου τμήματος της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Άρα φτάνουμε σε ένα σύνολο 32,3 δις. Αν δούμε λιγάκι την περιφερειακή κατανομή ε, υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα επιπρόσθετα 3 δις που ήταν μια ε, επιπρόσθετη δυνατότητα και τα 2,3 που προσθέτηκαν. Τα έξτρα 3 δι ε, ευρώ μοιράζονται, κατανέμονται σε 1,4 Αυτά αφορούν 900 εκατομμύρια της χώρας Μεσογείου και 500 εκατομμύρια ως προενταξιακή βοήθεια. Τα 1,2 δις αφορούν την Ανατολική Ευρώπη και κατανέμονται από αυτά αναλογικά σε όλες τις περιοχές. Αν δείτε λιγάκι αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχουμε 440 ε, εκατομμύρια με τη μορφή προενταξιακής βοήθειας και 1,86 δις στις χώρες της Μεσογείου. Αυτό ε, ίσως αυτή η δεν μπορείτε να τη διαβάσετε καλά, αλλά αυτό που αναφέρει είναι ότι υπάρχει κάποια αλλαγή. Δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην ε, Ανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Επίσης, επιφέρουμε και κάποιες άλλες αλλαγές στην πρότασή μας. Η πρώτη έχει σχέση με την κάλυψη σε σύνολο χώρας. Δηλαδή, Προτείνουμε να αφαιρεθούν από τον κατάλογο πλούσιες χώρες οι οποίες ε, βρίσκονται σε μια κατάσταση ε, που είναι παρεμφερής με τα κράτη-μέλη μας. Δηλαδή Μπρουνέι, Ισλανδία, Ισραήλ, Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα, Χονγκ και Μακάο. Επίσης ε, προτείνουμε μετά τα από πρόθεση της κυρίας Μογκερίνη να προσθεθεί το Ιράν στον κατάλογο των ενδεχομένως επιλέξιμων χωρών με μια διευκρίνηση. Αυτή η προσθήκη δεν αλλάζει όμως τίποτα. Δηλαδή το να γίνει το Ιράν επιλέξιμη χώρα, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει κατεξουσιοδότηση πράξης της Κομισιόν και εκεί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν δώσει τη δυνατότητα να διαφωνήσουν αν δεν συμφωνούν με αυτή την πρόταση. Άρα δηλαδή σε αυτή τη φάση αυτή η πρόταση είναι συμβολική, δεν είναι ουσιαστική, όμως η Αντιπρόεδρος κυρία Μογκερίνη ε, πιστεύει ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες συμβολικές κινήσεις έναντι του Ιράν μετά από τη συμφωνία που έχει προκύψει για να επιβραβευτούν οι προσπάθειές τους. Άλλη μεγάλη αλλαγή, μεγαλύτερη ευελιξία. Προτείνουμε ε, να αυξηθούν κατά 20% ε, τα κονδύλια που μπορούν να κατανεμηθούν γεωγραφικά εκτός από αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που αναφέραμε προηγουμένως γιατί για αυτήν ειδικά είχαν προβλεφθεί συγκεκριμένα ποσά είχαν προσημειωθεί ποσά. Πόσο κοστίζουν τώρα όλα αυτά. Αν θυμάστε, το ELM δουλεύει με το Ταμείο Εγγύσεων εμπροστοβαρός και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξηγήσουμε τις επιπτώσεις οι οποίες επιπτώσεις αναμένεται να είναι της τάξης των περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα δηλαδή προτείνουμε για πρώτη φορά να συσταθεί μία μορφή εσόδων για το Ταμείο Εγγύησεων, δηλαδή, δηλαδή μία νέα εγγύηση που τα αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Ε, μπορούμε να πούμε ας πούμε ότι αυτό τα κονδύλια θα διοχετεύονται στο Ταμείο Εγγύσεων όπως συμβαίνει και με το Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων. Και αυτό για να δείξουμε ότι υπάρχει κάποια προστασία του ε, προϋπολογισμού, μία προστασία που είναι σε αναλογία με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Τώρα πάμε στον κατάλογο που δείχνει το προβλεπόμενο δημοσιονομικό κόστος. πιστοβαρής είναι ο, ε, ο υπολογισμός. Προς το τέλος θα προκύψει δηλαδή το βάρος. Ας πάμε τώρα στον επόμενο κανονισμό όπου προτείνουμε κάποιες αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή είναι εκείνη που σας ανέφερα προηγουμένως, ότι υπάρχουν νέα έσοδα που θα διοχετεύονται στο Ταμείο Εγγύησεων. Η δεύτερη αλλαγή είναι μια μικρή αλλαγή ε, στο κατόφλι. Ε, πέρα από αυτό, τα ε, κονδύλια επιστρέφονται στα κράτη-μέλη. Ισχύει το ίδιο ανώτατο όριο για το Ταμείο Εγγύησεων όμως ε, επειδή αντιμετωπίζουμε νέους κινδύνους και επειδή υπάρχουν και νέες πηγές εσόντων, πρέπει ε, να υπάρχει δυνατότητα αυτά τα έσοδα να μπαίνουν σε ένα είδος ε, μαξιλαριού έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι επιπρόσθετοι κίνδυνοι που σήμερα όμως αυτοί δεν μπορούν να προβλεφθούν αυτό νομίζω ότι το γνωρίζουν όλοι και γι' αυτό το λόγο εμείς προτείνουμε ε, τα χρήματα να μην επιστρέφονται στα κράτη-μέλη όσο το ε, Ταμείο Εγγύσεων δεν φτάνει στο 10%. Δηλαδή παραμένουμε στην αρχή ότι ισχύει αυτό το 10%. Εάν τα ε, επιπρόσθετα έσοδα είναι κάπου στο 9 μέχρι 10%, ε, μέχρι το 10 δεν επιστρέφονται τα κονδύλια στα κράτη-μέλη για να υπάρχει καλύτερη προστασία του προϋπολογισμού. Αυτό είναι σημαντικό να το έχει κανείς κατά νου, γιατί το Ταμείο Εγγυήσεων καλύπτει επίσης και την ε, μακροοικονομική βοήθεια ε, το μέγεθος της βοήθειας έχει αυξηθεί, είναι τώρα πολύ μεγαλύτερη λόγω της Ουκρανίας και επειδή πρόκειται για μια γεωγραφική περιοχή όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ιδιαίτερα ενεργή, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι και ως εκ τούτου πρέπει αυτοί να ληφθούν υπόψη για να προστατεύεται καλύτερα ο ενωσιακός προϋπολογισμός. Η τελευταία αλλαγή την οποία προτείνουμε και είναι περισσότερο τεχνικής φύσεως είναι η διαχείριση κονδυλήσεων του Ταμείου Εγγύησεων που σήμερα έχει ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επανέλθει αυτή η διαχείριση στην ίδια για την Επιτροπή. Σήμερα έχουμε ποσά που μοιάζουν με αυτά που ε, διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χάρη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τα επόμενα έτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαχειρίζεται περίπου τα δύο τρίτα των κονδυλίων που έχουν τα διάφορα ταμεία και υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα οικονομίας κλίμακος. Άρα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προβαίνει στην διαχείριση των κοντιλίων χωρίς επιπρόσθετη πρόσληψη προσωπικού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι το κόστος της διαχείρισης των κοντιλίων αφαιρείται από το Ταμείο των Εγγύσεων που σημαίνει εξοικονομήσεις στις οποίες προβαίνουμε μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερα τόσο για το ELM όσο και για την μακροοικονομία οικονομική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Οι αποδόσει τη είναι περίπου ίδιε όπω και αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτρέπεται εξοικονόμηση περίπου ενό εκατομμυρίου ευρώ τον χρόνο. Μιλάμε για συνολικά 44 εκατομμύρια που φτάνουν μέχρι και τα 66 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι κριτική προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Απλά υπάρχει, όπως σας είπα, η δυνατότητα να επιτυγχάνουμε οικονομίες κλίμακος. Και εδώ σταματά την παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αγγέλ. Ήσασταν απόλυτα σαφείς. Δηλαδή έχουμε επιπλέον μια δυνατότητα τριών δις χρηματοδότησης. Και το 10-11% θα πρέπει να είναι από τον προπολογισμό και να τεθεί στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχουμε τρία δις που ήδη προβλέπονται, λέει ο κ. Σανζέλ, όπως ε, ως δυνατότητα στην απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και επειδή έχουμε τη νέα αίτηση για τους πρόσφυγες για την οποία η Τράπεζα Επενδύσεων εργάστηκε πάρα πολύ γρήγορα για να κάνει πρόταση έχουμε μια επιπλέον πρόταση 2,4 πέρα από τα 3 που θα επιτρέψει στην Τράπεζα Επενδύσεων να προτείνει καινοτόμες ενέργειες ε, που θα στρέφονται προς τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε πρέπει να καλυφθεί αυτό στον προπολογισμό και είναι 9% του συνολικού ύψους των, των ε, δανείων του στο έτος ε, νη 2. Δηλαδή θα εμφανιστεί αυτό το κόστος ε, κατά την διάρκεια της εξέλιξης των ε, δαπανών. Μένουμε λοιπόν στο 9% αλλά έχουμε και ένα περιθώριο ασφάλειας για τις νέες αυτές δραστηριότητε για να προστατεύσουμε τον προπολογισμό και να μην χρειαστεί να ζητήσουμε πλέον πόρους ενώ ένα τμήμα ε, των εσόδων θα έχει επανέλθει στον, στα κράτη-μέλη. Για τους πρόσφυγες, ναι, για τους πρόσφυγες. Και πού θα μείνουν αυτοί οι πρόσφυγες. Και στις χώρες όπου βρίσκονται, α όχι, πρώτα απ' όλα στις χώρες προέλευσης και στις χώρες προορισμού γιατί γίνονται κάποιες ενέργειες για όλες τις χώρες. Πρόεδρος. Και τι είναι ένας πρόσφυγας που μένει στη χώρα προέλευσής του. Νο, όχι, όχι, στις ε, περιοχές προέλευσης. Στις ζώνες προέλευσης. Στην Ιορδανία για παράδειγμα και την Τουρκία. Στην Ιορδανία για παράδειγμα έχουμε. Έχουμε περίπου ένα εκατομμύριο πρόσφυγες όσα μπορεί να κάνει η ΕΤΕ για να βοηθήσει στην Ιορδανία για να υπάρχει απασχόληση, να υπάρχουν υπηρεσίες για αυτούς τους πρόσφυγες. Όλα αυτά θα βοηθήσουν οι πρόσφυγες αυτοί να μην φύγουν και να μην έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πω πιο απλά, πιο αδρά. Πρόεδρος, βλέπουμε όλοι αυτό το μηχανισμό, αυτά τα δισεκατομμύρια αλλά ποια είναι η συνολική σας προσέγγιση. Ποια είναι η στρατηγική σας, η γενική στρατηγική σας. Ποια είναι η μακροπρόθεσμη προοπτική. Το 2050 η Αφρική θα έχει 2 δισεκατομμύρια κατοίκους. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, λέει ο κύριο Σανζέλ, πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η εξωτερική εντολή, που είναι κάτι που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Η πάντα είχε τέτοιες εξωτερικές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα υψηλέ οι πρικοδοτήσεις του οι προκοδοτήσεις της αυτής εντολής. Υπάρχει το νέο ταμείο, αυτό το EFSD, που θα πάρει 1,5 εκατομμύριο για Δηλαδή είναι 5 επιπλέον των 27, δηλαδή είναι πολύ σημαντικά ποσά για τα οποία η ΕΤΕ έχει ήδη μεγάλη πείρα, ένα μεγάλο τμήμα της δραστηριότητας ΕΛΜ έχει να κάνει με την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί η ΕΤΕ να ανταποκριθεί καλύτερα στα αιτήματα που έχουν ε, υποβληθεί από τις ανώτατες πολιτικές αργέ να αναπτύξει δραστηριότητες που δεν έκανε πριν. Ποιο είναι το πιο υψηλό επίπεδο, αργή κρατών και κυβερνήσεων. Τον περασμένο Μάρτιο κάλεσαν την ΕΤΕ να αναπτύξει πρωτοβουλίες. Γι' αυτό το στόχο. Και αυτό έκανε η ΕΤΕ. Πρόεδρος. Ναι, αλλά θα θέλαμε να εκφραστεί μια πολιτική προσέγγιση. Θα μας πούνε αρχή κρατών κυβερνήσεων ποιος είναι ο στόχος τους. Κύριε Πρόεδρε, λέγομαι Ρομπέρτο Ριντόφι από την ΤΕΦΚΟ. Είναι το επόμενο σημείο, αλλά να παρέμβω τότε. Για να σας ε, δώσω επιπλέον στοιχεία. Η ανακοίνωση του Προέδρου της 14ης Σεπτεμβρίου, στην οποία παρουσιάζεται το πρόγραμμα εξωτερικών επενδύσεων. Αυτή, αυτό είναι το όραμα. Δεν υπάρχει βιώσιμη λύση εάν δεν αποφασίσουμε να επενδύσουμε περισσότερο για να υπάρξει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Αφρική. Έτσι λοιπόν συνδυάζουμε διάφορες δυνατότητες για να εξυπηρετήσουμε αυτήν την προοπτική, να υπάρξουν επενδύσεις, για να υπάρξει απασχόληση, Αυτό θέλω τώρα να σας παρουσιάσω. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την ε, πρόσκλησή σας. Και σας ευχαριστώ πολύ. Τον Ιούνιο είχαμε μια ανακοίνωση για τη νέα εταιρική σχέση. Για μια προσέγγιση πλαίσιο που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι φιλόδοξο. Στις 14 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος Γιούνκερ έδωσε αυτή τη φιλόδοξη προσέγγιση. Ο στόχος του είναι να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ και παράλληλα να αντιμετωπίσει τις βασικές αιτίες της οικονομικής μετανάστευσης. Δεν εξετάζουμε τα θέματα σειράξεων, αν και θεωρούμε ότι αν υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη θα μειωθούν τα αίτια σειράξεων σε πάρα πολλές χώρες. Αλλά η οικονομική μετανάστευση είναι αυτή που προκαλείται από την ένδυα. Γι' αυτό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μικρό τμήμα των πιστώσεων αυτών από ότι είναι διαθέσιμα στα, στο πολιτές πλαίσιο με τρόπο που να μοχλεύσουμε πολύ υψηλές επενδύσεις όχι μόνο από τους συνήθεις υπόπτους στην ΕΤΕ, αλλά και από τις ε, κανονικές ε, τράπεζες, την Κάσα Ντεπόστα στην Ιταλία, την ΚΕΒΕ, την Κοφίντε στην Ισπανία και άλλες, αλλά και από ιδιωτικές επενδύσεις. Τα 3 εκατομμύρια που κάθονται στα συνταξιοδοτικά ταμεία που και δεν καταφέραμε να κινητοποιήσουμε μέχρι στιγμή για να επενδύσουν στις τρίτες χώρες. Γιατί δεν επενδύουν στις τρίτες χώρες, γιατί οι κίνδυνοι που βλέπουν οι διοικητέ των ταμείων αυτών είναι πολύ ψηλή. Και δεν είναι μόνο έτσι η, η εντύπωση που έχουν, γιατί και εγώ έχω ζήσει 15 χρόνια στην Αφρική ω πρέσβη τη Ένωση και πρέπει να σα πω ότι η κίνδυνη είναι πραγματική. μη τάξη, διακυβέρνηση, υπάρχουν πολιτικά θέματα, διαφθορά. Αλλά από οικονομική πλευρά υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που θέλει να αντιμετωπίσει η Κομισιόν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης που αποτελείται από τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι μια πρόταση επενδύσεων με καινοτόμες εγγυήσεις 1,5 δις επιπλέον. Επιπλέον δύναμη πυρός. Αλλά για να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτησή σας, κύριε Πρόεδρε, συνδυάζοντας τα ταμεία του αναπτυξιακού ταμείου, με τα χρήματα του αναπτυξιακού ταμείου, με τα χρήματα του προπολογισμού, έχουμε περισσότερη δυνατότητα λογοδοσία προ το κοινοβούλιο και ελέγχου από το κοινοβούλιο. Και έχουμε και από το αποσματικό του EDF 400 εκατομμύρια του αναπτυξιακού ταμείου, που επίση θα αξιοποιήσουμε, καθώς και κάποια χρήματα από το ENI, που θα είναι πόροι του προπολογισμού και άρα θα ελέγχονται από το Κοινοβούλιο. Συνδυάζοντα λοιπόν πόρους του Αναπτυξιακού Ταμείου και του προπολογισμού, αυξάνουμε το επίπεδο λογοδοσίας ε, της Κομισιόν. Το δε, η δεύτερη συνιστόσα του πυλώνα, του επενδύσεων είναι η δυνατότητα συνδυασμού περιφερειών. Το κάνουμε εδώ και κάποια χρόνια αυτό, αλλά θέλουμε να το κάνουμε περισσότερο, για να υπάρχει περισσότερο συντονισμό και με άλλε δράσει πολιτική και άλλε πολιτικέ. Σε αυτά που κάνουμε εκτό Ένωση. Αναφερθήκατε στο ΕΦΣΙ, κύριε Πρόεδρε. Από πλευρά μόχλευση, βεβαίω είναι παρόμοιοι συντελεστέ. Αλλά οι ομοιότητε ε, είναι επιφανειακέ. Γιατί Πολύ συχνά εμείς δρούμε σε ένα εχθρικό περιβάλλον, σε χώρες εταίρους, όπου υπάρχουν αρκετές ελλείψεις. Δεύτερον, γιατί οι στόχοι πολιτικής που έχουμε πρέπει επίσης να γίνουν σεβαστοί. Οι κανονισμοί, το ENI, το DCI, από όπου έρχονται τα χρήματα. Και βεβαίως και το Αναπτυξιακό Ταμείο. Πρέπει να σεβαστούμε τους στόχους πολιτικής, επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία αυτών των μέσων. Έχουμε λοιπόν πολιτικές ευθύνες και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε για τις ίδιες αρχές χρηματοπιστωτικής μόχλευσης που χρησιμοποιούμε επιτυχημένα για το ΕΦΣΥ. <clears throat> λοιπόν, ο δεύτερος ε, πυλώνας είναι 4,1 δις, είναι αυτός ο χρηματοδοτικός μηχανισμός και ο άλλος πυλώνα είναι η τεχνική βοήθεια. Γιατί ξέρετε, πολύ συχνά υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση, αλλά δεν υπάρχουν προγράμματα που να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Άρα πρέπει και οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτήσεις όχι μόνο από την Ένωση αλλά και από ιδιωτικούς επενδυτές. Αυτοί έχουν τα 3 εκατομμύρια που λόγω της σημερινής οικονομικής κατάστασης δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Οπότε, τεχνική βοήθεια για να τους βοηθήσουμε να μπορέσουν να πάρουν χρηματοδοτήσεις. Και τρίτον, να υπάρχει ένα ε, δομημένο διάλογο με τι κυβερνήσει, με τι επιχειρήσει, για να βελτιωθεί η ανομή τάξη, για να καταλάβουν ποια είναι τα κριτήρια επενδύσεων, για να υπάρχει νομοθεσία που να προστατεύει τι ξένε επενδύσει. Ο πυλώνας αυτό είναι επίση πολύ σημαντικό. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι δουλεύουμε και για τους τρεις αυτούς πυλώνες με πολύ καινοτόμο τρόπο, από κοινού, δημιουργώντας ένα ταμείο εγγύσεων για τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει να επενδύσει το εξωτερικό ταμείο, ε, πρόγραμμα επενδύσεων, θα ασχοληθεί με κοινωνικές υποδομές, θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες για να δημιουργήσουν απασχόληση. Λόγω των σημερινών δημογραφικών τάσεων που σημαίνουν ότι πρέπει να δημιουργηθούν 18 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας το χρόνο μέχρι το 2035 στην Αφρική και μάλιστα να είναι αξιοπρεπείς και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Επιμένω, αξιοπρεπείς και βιώσιμες. θέλουμε ε, να γίνουν η Κίνα μας αυτή. Αν δούμε τι κάνει η Κίνα σε πολλές αφρικανικές χώρες, θέλουμε και εμείς να κάνουμε αυτό. Κάνει τρομερές επενδύσεις. Χωρίς καμία διαφάνεια, χωρίς καμία βιωσιμότητα, χωρίς καμία αξιοπρέπεια, χωρίς καμία ε, φροντίδα για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Αλλά το κάνουν. Είναι τεράστιες επενδύσεις. Αξιο... Ε, εντυπωσιακέ. Και επίσης, να τονίσω τα εξή. Η διακυβέρνηση που θα βασιστεί με αυτή τη δυνατότητα συνδυασμού πόρων είναι κάτι επί το οποίο εργαζόμεθα με το 2008. Μας έχουν δώσει πολύ, καλή, ε, πολύ καλά αποτελέσματα γιατί όχι μόνο εργαζόμεθα με πολύ καλές υπηρεσίες της ΕΤΕ αλλά και με κάποιους άλλους. Πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Πολύ περισσότεροι πρέπει να κινητοποιηθούν για να επιτύχουμε αυτά τα νέα αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής Κατά την περίοδο 2007-2015 η Ένωση έχει δώσει 2,7 δις αυτές τις συνδυασμένες επιχειρήσεις που κινητοποίησαν πόρους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 23 δις για να στηρίξουν 278 προγράμματα, συνολικός προϋπολογισμός 50 δις. Νομίζω τα στοιχεία αυτά τα αναφέραμε πρόσφατα όταν κάναμε τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου με βάση τις συστάσεις του οποίου που καλούσαν για περισσότερη προσθετικότητα, δηλαδή τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων να κινητοποιούν επενδύσεις, αλλιώς να μην χρησιμοποιούνται και όπως είπα και προηγουμένως πρέπει να διαχειριστούμε κινδύνους πολιτικής και πολιτικών. Η λογοδοσία είναι βασική έννοια για μας γιατί ετησίως έχουμε υποχρέωση να υποβάλουμε εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και το αναφέρει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και μια έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στον κανονισμό. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να διαχειρίζονται, να τις διαχειριζόμεθα με βάση και τις πολιτικές της ε, ΕΤΕ. Μαζί και με την Τράπεζα Βιώσιμη Ανάπτυξη, με το Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξη, όλα αυτά είναι όργανα τη εξωτερική μα πολιτική στα πλαίσια τη ευρύτερη πολιτική διαλόγου που κάνουμε με τι ε, χώρε εταίρου οι επενδύσεις δεν θα πιάσουν και δεν θα έχουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αν δεν υπάρχει αυτός ο πολιτικός διάλογος. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει αναλάβει πλήρως τη δίκηση αυτού του προγράμματος και επειδή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, είναι αρμόδια για το διάλογο αυτό, καλύπτουμε πλήρως το φάσμα, συμμετέχουν όλοι οι φορείς ακόμη και η μη ενωσιακή. Για παράδειγμα, η Αφρικανική τράπεζα, Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι βασικός παράγον. Ο ρόλος της ΕΤΕ θα ενισχυθεί στα πλαίσια αυτά. Προτείναμε να είναι μέλος του Στρατηγικού Ταμείου του Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης και να είναι τεχνικό σύμβουλος για τη γραμματεία του Ταμείου αυτού για τη διαχείριση των εγγύσεων από χρηματοοικονομικής πλευράς, αλλά θα είναι και βασικός εταίρος μας στην προσπάθεια εκτέλεση των προγραμμάτων. Καταλήγοντας, η Επιτροπή είναι σε πολύ κατάλληλη θέση για να λάβει την ευθύνη για τη διαχείριση και του, της ΕΤΕ και του Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω των τριών πυλώνων και των διαφόρων πλευρών του διαλόγου και για να λάβει την πολιτική ευθύνη. Έχει και την συνολική επισκόπηση και τις αναγκαίες πιστώσει. Έχουμε διάφορα μέσα, ορισμένα ήδη τα αξιοποιεί η Κομισιόν και είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε την ε, συνοχή όλων των εξωτερικών δράσεων. Αυτό το Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν ξεκινάει εν κενό. Υπάρχει μια πληθώρα άλλων πρωτοβουλειών και δημιουργία λοιπόν μιας πύλης, μιας ε, ενιαίας στηρίδας για να απευθύνονται όσοι θέλουν να κάνουν επενδύσεις μια προσέγγιση δηλαδή φιλική προς τον χρήστη, προς τον πελάτη είναι πολύ χρήσιμη. Η Κομισιόν βεβαίως ε, λογοδοτεί έναντι του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρα πρέπει να διοικεί και να αναλαμβάνει ευθύνε και θα διασφαλίσουμε και την προστατικότητα, θα, εστιάσουμε στην μείωση της φτώχειας και την επίτευξη αξίας, ε, προστιθέμενης αξίας. Ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις διευκρινήσεις. Ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε στο μόνιμο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις Βρυξέλλες να μας πει πώς τα βλέπει όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα τα πω αγγλικά και υπόσχομαι να είμαι λακωνικός διότι είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και ερωτήσεις. Τους τελευταίους δύο μήνες ε, κάναμε πολλά πράγματα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και το ELM, το ε, ε, εξωτερικό δανεισμό την εντολή εξωτερικού δανεισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων και συνεργασία ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη και να συμπληρώνουμε απλώ ένα τον άλλον. Και αυτό μας το ζητά συνεχώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διάφοροι πολιτικοί φορέ στο Συμβούλιο και είμαι σχεδόν βέβαιο ότι θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Δεν νομίζω ότι ε, μπορεί να γίνει και αλλιώ άλλωστε. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει πολύ καλό ε, ιστορικό όσον αφορά την τεχνική της εμπειρογνωμοσύνη αλλά και την αποτελεσματικότητα από πλευράς προϋπολογισμού των διαφόρων μέσων που υλοποίησαμε. Το 2015 δώσαμε περίπου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ δανειοδότησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 55% αυτού του ποσού έγινε βάσει τη εντολής ε, εξωτερικού λεδανισμού 30% στον ίδιο κίνδυνο και ε, το υπόλοιπο ποσοστό ε, δανεισμός βάσει της συμφωνίας του Κοτονού. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουμε επιπλέον ε, επίπεδα γραφειοκρατίας, να μην υπάρχει επικάλυψη των κυβερνητικών δομών και καθεξής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των μέσων με την ε, δυνατότητα επενδύσεων και την εντολετική εξωτερικού δανεισμού και αυτή τη νέα πρωτοβουλία ε, της Ευρωπαϊκής Τραπέζας ε, Επενδύσεων για την προσαρμοστικότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τα όσα έχουμε προβλέψει στα υπάρχοντα μέσα. Θα ήθελα να πω το εξή για την εντολή εξωτερικού Ευχαριστούμε βέβαια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ό,τι έκανε προκειμένου να βρει περιθώριο να ε, ε υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία προσαρμοστικότητας ε, βάσει των όσων αποφασίστηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι δύσκολη η πολιτική πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να σας το αναφέρω αυτό διότι ακόμα και με την αύξηση στην εντολή εξωτερικού δανεισμού θα υπάρχει σημαντική μείωση του δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κυρίως στην Ανατολική Γειτονία, θα μειωθεί κατά 70% σε σύγκρουση με τα τρέχοντα επίπεδα. Επίσης θα υπάρχει οξύτατη μείωση στην Ασία, στη Λατινική Αμερική και την Νότια Αφρική, ε, περίπου 50% και μιας και αναφέρθηκε και το Ιράν, ε, και άλλες ε, δυνητικές νέες χώρες, Λευκορωσία, Μιανμάρ, ε, Κούβα, τις ανέφερε ο Μπένζαμιν. Θα πρέπει να είμαι σαφής εδώ, δεν έχουμε λεφτά να δοθούν για επιχειρήσεις σε αυτές τις χώρες. Έτσι έχει η κατάσταση. Κατανοώ βεβαίως ότι υπάρχουν πιέσεις στον προπολογισμό και περιορισμοί. Εδώ συζητάμε 34 εκατομμύρια μέχρι το 2020 και από εκεί και πέρα 165 για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό είναι το απαραίτητο ποσό ώστε να μπορέσει να δοθεί 6,2 δις δανειοδότηση επιπλέον από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να έχουμε τα επίπεδα που έχουμε και τώρα στην ε, Ανατολική Ευρώπη, στην Ασία, στην Νότια Αφρική. Ε, και στη Λατινική Αμερική. Ε, ξέρω ότι δεν είμαστε Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, επομένως ε, δεν θα επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες και το πόσο σημαντικό είναι αυτό αυτή τη στιγμή δεδομένων των συνθήκων, αλλά είμαι υποχρεωμένο να σας το αναφέρω εδώ και ελπίζω ότι παρά το γεγονός ότι πρέπει να είμαι ρεαλιστή και ξέρω ότι είναι δύσκολη συζήτηση όταν πρόκειται για προπολογισμό, θα το συνεχίσουμε να το αναφέρουμε το σημείο αυτό σε διάφορα επίπεδα στο Συμβούλιο και ήθελα να το θέσω και εδώ υπόψη σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν. Να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους που επιθυμούν να το λάβουν. Ο κύριος Ντονανό και μετά ο κύριος Δεπρέ. Κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να τα επεξεργαστούμε τα θέματα αυτά, διότι έτσι η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο στο σημερινό κόσμο, που είναι και όλο ένα και πιο σημαντικό, και επομένω στον προπολογισμό μα θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τον τίτλο 4 και ό,τι μπορεί να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει. Το Ευρωπαϊκό αυτό Ταμείο λοιπόν Βιώσιμης ανάπτυξη που θα συσταθεί ε, θεωρώ ότι αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση. Η κατάσταση σήμερα μας υποχρεώνει ουσιαστικά να δράσουμε. Με την παρέμβαση της Κίνας, ε, για παράδειγμα, και την περίπτωση της ε, ε, Αφρικής, ξέρω πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Ξέρω ότι η Κίνα είναι παρούσα. Και ξέρετε, ο πρόεδρος, τι διαφορά υπάρχει μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί έχουν λεφτά. Ε, δεν είναι το ίδιο. Ναι, έχουν λεφτά, επομένω είναι πανταχού παρόντε. Ε, υπάρχουν και άλλε χώρε που έχουν χρήματα. Ε, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεδομένων και των αποτελεσμάτων των εκλογών σήμερα, αλλά θα υπάρχουν ε, επιρροέ στην Αφρική και πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα στην Αφρική για να βοηθήσει στην ανάπτυξή τη, να βοηθήσει επίση και του Αφρικανού πολίτε να ζουν και να εργάζονται στην ήπειρό τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένων και των θεμάτων τη μετανάστευση που υφέρπουν. Επομένως, το Ταμείο συστήνεται και γι' αυτό, αλλά και για να βοηθήσουμε του πρόσφυγες που ήδη έχουν εγκατασταθεί σε κάποιες χώρε. Θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα, αλλά έχει τις ίδιες αδυναμίες με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι φτιαγμένο στο ίδιο μοντέλο, βασίζεται σε κάποιες εγγυήσει, Επομένω έχει και τι ίδιε αδυναμίε. Δεν υπάρχει φρέσκο χρήμα, δεν υπάρχει δημόσιο χρήμα και νομίζω ότι από εκεί ε, περιμένουμε από αυτούς τους κανόνες να έχουμε μόχλευση. Υπάρχει βέβαια και υπό όρους ε, δυνατότητα, αλλά αν πιστεύω ότι αν κάνουμε μια επιπλέον προσπάθεια ε, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε και τη μόχλευση. Και επίσης Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων υπάρχουν κάποιοι επιπλέον περιορισμοί για την Αφρική και νομίζω ότι τις επεσήμαναν οι ομιλητές. Αυτό που θα ήθελα να πω σήμερα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι παρόν για τα θέματα αυτά. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει κάπου πάρει τα ενία και εγώ ναι δεν θέλω να υλοποιήσει τα, τα όσα είπε, να αναλάβει την εκτέλεση και τη διαχείριση, αλλά θα ήθελα και να προσθέσουμε κάπου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λόγο, κυρίως όσον αφορά τους προσανατολισμούς και νομίζω ότι θα υπάρχουν και εγγυήσει και θα πρέπει να μιλήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και να υπενθυμίσω ότι είμαστε συνομοθέτες. Υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία αδυναμία και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το είπατε και εσεί, κύριε Πρόεδρε και πρέπει να επιμείνουμε από αυτού. Ε, θα λέει το άρθρο 15 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ε, ετήσια έκθεση και θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι αρκεί αυτό. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί περισσότερο και θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο και θα επιτρέψει και στην Ευρώπη να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο της ε, και να βοηθά στην ε, παρουσία της ανά τον κόσμο αλλά και στην ανάπτυξη της Αφρικανικής Υπήρου και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε να έχει και ένα πιο βέβαιο μέλλον η Αφρική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με το σύστημα εγγυήσεων και με το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τόσο έλεγχο. Ευχαριστώ κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είμαι η Δήμον σε θέματα εξωτερικών σχέσεων ούτε χρηματοπιστωτικών μέσων. Τώρα όλα αυτά τα ΕΝΗ, e, το SSD, το LLM, όλα αυτά και τις κάπως ανόμιες ε, παρουσιάσεις που μας κάνατε. Αυτό το νέο μέσο που μας παρουσιάζεται, πάντα θεωρούσα, εκτός αν κάνω λάθος, ότι σχετίζεται με, στο, με το στόχο του ελέγχου της μετανάστευσης. Το διάβασα αυτό. Το υπενθύμησε ένας από τους ομιλητές ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί να δημιουργηθούν με κάθε χρόνο 18 εκατομμύρια θέσουν εργασία. Αυτό μας είπατε. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξή. Σε σχέση με αυτό το στόχο, να σταματήσουμε την αναχώρηση των ενδεχομένων μεταναστών. Τι επιπλέον προσφέρει για το στόχο αυτό και σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση αυτή η νέα πρωτοβουλία σε μια περίοδο ετήσια ή μέχρι το 20. Πού θα τα κάνετε αυτά. Έχετε προσδιορίσει πού θα γίνουν αυτές οι δραστηριότητες, υποθέτω. Και τρίτον, πόσα θα μας κοστίσει εάν έπρεπε να το χρηματοδοτήσουμε για μία επταετή περίοδο που είναι η περίοδος των πολιετών προοπτικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να κάνω και εγώ μερικές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, για το Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης το ποσοστό μόχλευση είναι 12, ο συντελεστής μόχλευσης, ενώ για το ΕΦΣΙ είναι 15. Είμαστε στην Αφρική. Σε χώρε που για τους επενδυτές ε, είναι πολύ σχετική η ασφάλεια. Συντελεστή μόχλευσης 12. Σας φαίνεται λογικό. Γιατί η εγγύηση εντάξει, βάζουμε 9% στον κουμπαρά. Αλλά αν μετά προκύψουν προβλήματα, το 9% δεν τα καλύπτει. Θα τα χάσετε όλα όσα έχετε επενδύσει. Θα ήθελα να μου πείτε γιατί θεωρείτε ότι είναι καλός αυτός ο συντελεστής 12. Πρώτη επιφύλαξη. Η κυρία Γαρδιαθάμπαλ που ήθελε να είναι εδώ αλλά χρειάστηκε να φύγει είχε ερωτήσεις τις οποίες θα προσπαθήσω να σας θέσω εκ μέρους της. Ήθελε να μας πείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των προγραμμάτων που υποφελούνται από την εγγύηση του Ταμείου αυτού των προγραμμάτων που θα γίνουν ε, στα, πλαίσια τους, της διευκόλυνσης ε, για την Αφρική και ε, τα προγράμματα μέσω του προγράμματος επενδύσεων της ΕΤΕ. Σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις, γιατί αν πρέπει να εξηγήσουμε στους συναδέλφους πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά, θα είχαμε κάποιες δυσχέρειες. θέλαμε λοιπόν μια συνολικότερη προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα γεωγραφικά, μετά με ποιους στόχους και τέλος κύριε Φρέζα. Όλα αυτά ε, είναι συμβατά με το ισχύον πολιτές πλαίσιο ή θα χρειαζόταν μια αναθεώρησή του. Γιατί ξέρετε ανακυκλώνουμε κάτι μικροποσά που βρίσκουμε εδώ, βρίσκουμε από εκεί. Παίρνουμε από το αναπτυξιακό ταμείο που δεν ελέγχουμε καθόλου εμείς. Και μετά παρακαλάμε τα κράτη-μέλη να δώσουν κάτι και δεν ξέρουμε αν θα δώσουν. Δεν είναι λίγο περισσότερο διακηρύξεις όλα αυτά, ε. έτσι, τελετουργικές. Και λιγότερο ένα αξιόπιστο σύστημα που ξεκινάει με καθορισμένες ε, γεωγραφικές προτεραιότητες και προσπαθεί να επιτύχει συγκεκριμένου στόχους γιατί αν πάει κανεί επί τόπου δεν είναι προφανές πόσο βλέπει κανείς τι κάνει η Ευρώπη γιατί περνάμε από την Ηνωμένα Έθνη και πολλού άλλου εξωτερικού οργανισμού καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι η Ευρώπη είναι άλλη μία μη καπαόμικρον. Κλείνω την παρένθεση. Είναι μία συζήτηση που σίγουρα συγκινεί πάρα πολύ τους παρευρισκόμενους γιατί μίλησαν όλοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για να απαντήσω στις τελευταίες σας ερωτήσεις. Ε, αν αυτά τα οποία προτείνονται συνάδουν με το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο ε, ή όχι. Ναι, είναι συμβατά και αυτό βασίζεται και στις προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Επομένως χρειάζεται μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Ναι, είναι στη δέσμη των μέτρων της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης ένα μεγάλο τμήμα, τα 250 επιπλέον εκατομμύρια, αυτό του φρέσκου χρήματος αν θέλετε, για το Ταμείο Εκκοιήσεων, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι στη διορθωτική επιστολή του προπολογισμού του 2017. Χωρίς δηλαδή την διορθωτική επιστολή υπαριθμών 1 δεν έχουμε τίποτα. Ναι, ακριβώς. Θα χρειαστεί να υπάρξει συμφωνία λοιπόν επ' αυτή τη βάση στον προπολογισμό. Για ε, τα κονδύλια λοιπόν ε, που προβλέπονται είναι αυτά τα, ε, θα παραμείνουν και είπαμε θα έχουμε τη διορθωτική επιστολή και θα έχουμε και 25 εκατομμύρια που θα είναι από το μέσο γειτονία. Αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και πρέπει να υπάρξει μετά συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 2017 βεβαίως. Και επίσης να πω ότι ε, στη δέσμη αυτών των προσθήκων που κάνουμε στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση θα έχουμε και αυτά τα 150 εκατομμύρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην εταιρική ε, σχέση μεταξύ τρίτων χωρών ή χωρών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποια μέτρα είτε σε οικονομικό επίπεδο είτε σε θέματα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών με τις χώρες εταίρους και εδώ έχουμε αυτά τα 150 εκατομμύρια τα οποία προβλέπονται και αυτά ε, και πάλι θα ε, συμπεριληφθούν στον προπολογισμό του 2017. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα οποία συνάδουν με το παρόν πλαίσιο και για το 2017 βάσει ε, και των συμφερόντων της Ένωσης και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα ελπίζουμε αυτές οι παράλληλες διαπραγματεύσεις που γίνουν, που ελπίζουμε να συγκλίνουν κάποια στιγμή για τον προπολογισμό του 2017 και την αναθεώρηση του πολιτού πλαισίου, θα μας οδηγήσουν σε μια αποδεκτή λύση ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Ε, επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Αντόλφη, ο οποίος θα απαντήσει στις άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την πρώτη Αναμφίβολα υπάρχει υποχρέωση να δράσουμε και θα ήθελα να απαντήσω και στο ερώτημα πόσο ε, θα μπορούσαμε να ορίσουμε αν θα ήταν για 7 χρόνια γιατί αντί για 3-4. Έχουμε εδώ το πρώτο καλό παράδειγμα για την εφαρμογή των νέων χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη. Αυτό συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2015 στην Αντίσα Μπέμπα. Και εκεί προβλέπεται μεγαλύτερη κινητοποίηση πόρων, έτσι ώστε οι χώρες αυτές να μπορούν να εφαρμόζουν φορολογία, αλλά και να εφαρμόζονται και αυτές οι δράσεις, δηλαδή τα χρήματα να μην χρησιμοποιούνται ως ενισχύσεις, δηλαδή να μην κατασκευάζεται ένα εργοστάσιο παραγωγής, παραγωγής ενέργειας, με ενισχύσεις δεν μπορούμε να μιλάμε για ε, δώρο αλλά για ε, κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η υποχρέωση δράσης που σημαίνει ότι στα 7 χρόνια θα πρέπει να επενδυθούν περισσότερα χρήματα. Και αυτή είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή. Όσον αφορά την αδυναμία του ΕΨΗ, του προγράμματος ε, των, της πρωτοβουλίας των στρατηγικών επενδύσεων. Ξέρουμε ότι η Κίνα έχει λεφτά, κύριε Πρόεδρε. Όμω, αυτά τα χρήματα συναντεύονται με ένα πολύ μεγάλο τίμα Όταν εγώ ήμουν πρέσβη στην Ογκάντα, ο πρόεδρος μου είχε πει θέλουμε να κάνουμε δουλειέ με τους Ευρωπαίους και όχι με του Κινέζους, αλλά εσεί δεν έρχεστε να μας κάνετε μία προσφορά. Αυτό λοιπόν το σχέδιο μα δίνει τη δυνατότητα να του απαντήσουμε θετικά ε, και να ε, συνοδεύσουμε τα χρήματα αυτά και με κάποιε αρχές που είναι σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν λέω ότι πρέπει να αναμίξουμε τα χρήματα του EDF με τα δημοσιονομικά κονδύλια, αυτός είναι και ο ρόλος που μπορεί να παίξει το Κοινοβούλιο οποτεδήποτε ε, αποδίδει στρατηγικό προσανατολισμό στον στρατηγικό μας προγραμματισμό. Θα υπάρξει ενδιάμεση αξιολόγηση ε, και αυτό που θα παίξει ρόλο είναι όχι τόσο τα κονδύλια όσο το πολιτικό στοιχείο. Και για να απαντήσω στην ερώτηση, ποιε είναι οι επιπτώσεις σε σχέση με τη δημιουργία τέσσεων απασχόληση για του χρόνου. Ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξης δεν προσποιείται ότι έχει βράχη πρόθεσμη απάντηση, αλλά μακροπρόθεσμη. Δημιουργούμε βάση για επενδύσεις που χρειαζονται δυο δύο-τρία χρόνια για να αναπτυχθούν περαιτέρω Επίση και άλλα τόσα χρόνια, γιατί έχουμε εμπειρία. Όταν κατασκευάζουμε, παραδείγματο χάρη, ένα δρόμο, οι επιπτώσεις, οι πραγματικές, προκύπτουν μετά από 5-6 χρόνια. Γι' αυτό, αν ρωτήσει κανείς ε, μέσα από αυτό το ε, ταμείο τι θα επιτύχει κανείς τα επόμενα τρία χρόνια, θα πω τίποτα. Όμως, η εμπιστοσύνη στους επενδυτές ότι αυτές οι δράσεις θα εμπνεύσουν αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε πολλές επενδύσεις να ξεπεράσουν το θέμα του κινδύνου. Και όσον αφορά την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν τα κονδύλια, θα ήθελα να πω το 80%, αν μιλάμε για το 80%, το 60% θα προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και πρέπει να επενδυθεί στην Αφρική αυτά που προέρχονται από το μέσο της γειτονίας θα πρέπει να επενδεθούν ε, στις χώρες προς Νότον και προς Ανατολάς. Προσπαθούμε λοιπόν να ε, σεβαστούμε και το γεωγραφικό στοιχείο. Και όσον αφορά στο θέμα του κινδύνου, κύριε Πρόεδρε, λέτε γιατί 11 και όχι 15. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι οι δουλειές που θέλουμε να δημιουργούμε κάθε χρόνο είναι 18, 18 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Και όσον αφορά τη μόχλεψη, προτείνουμε 11. Γιατί είναι πολύ πιο επικίνδυνο να επενδύσει κανείς στην Αφρική και γι' αυτό δεν μιλάμε για 15. Προτείνουμε όμως και κάλυψη της εγγύησης που είναι το 50% σε χρήμα, κινητοποίηση λοιπόν χρήματος για να καλυφθεί η εγγύηση, αντί για το 30-35% του ΕΦΣΥ. Και πάλι γιατί εδώ μιλάμε για μεγαλύτερο κίνδυνο. Μιλάμε λοιπόν ένα ποσοστό να, για την εγγύηση να κινητοποιηθεί με τη μορφή χρήματος και μικρότερη μόχλευση λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας του περιβάλλοντος. Και νομίζω ότι έτσι μπορώ και απαντώ στις ανησυχίες σας. Και ολοκληρώνοντας, όσον αφορά τη περίφημη αυτή μονοπευθυντική θηρίδα, γιατί έχουμε τρεις πυλώνες και όχι έναν, εμείς προτιθέμετα να εξορθολογήσουμε όλες τις ενέργειες που αναφέρθηκαν προηγουμένως υπό την ίδια προσέγγιση, έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση, αλλά ούτε και ανταγωνισμός ανάμεσα στις διαφορές πράξεις. Ε, πολύ σημαντική είναι διαφάνεια και υπάρχει κάτι που δεν το ανέφερα. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει στο να κινητοποιήσει κατά κάποιον τρόπο και τον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση που θα βοηθήσει όλους, θα βοηθήσει και τον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε και αυτός να επενδύσει στην Αφρική. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε όλο και περισσότερο στο μέλλον. Αυτά έκανα να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες αυτές και τη φιλόδοξη προσέγγισή σας, αλλά παρακαλώ να πείτε στους αργούς κρατών και θα το πούμε και εμείς ότι δεν πρέπει να υποτιμούν δεν πρέπει να υποτιμούν ε, τι πρόκληση θα αποτελέσει δημογραφικά η Αφρική. Και αυτά που μας προσφέρεται μπορεί να είναι εντυπωσιακά από πλευρά ύψου. Αλλά τα χρήματα που θα εγγυήσετε, που θα βάλετε ε, κατά μέρο για να εγγυηθείτε κάποια επένδυση, ακόμη και με 11 ε, συντελεστή, μου δημιουργεί κάποιες ανησυχίες. Σε μια χώρα, για παράδειγμα, όπως η Αργεντινή, όταν ο λαός αντιμετώπισε την απόλυτη ανέχεια, άρχισαν να μην πληρώνουν ε, τις κοινοφιλείς υπηρεσίες, ηλεκτρικό και νερό. Και βέβαια ένα εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να χτιστεί μόνο με επιδοτήσεις. Άρα δεν πρέπει να υποτιμούμε τις οικονομικές ανάγκες που θα χρειαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ για αυτό το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Κύριε Πρέζα, σας ευχαριστώ που μας δώσατε επιχειρήματα για να πείσουμε το Συμβούλιο για να ε, ε, καταλάβουν πώς πρέπει να γίνει η, ανα, η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Αν οι συνάδελφοι συμφωνούν, μπορούμε να κλείσουμε από αυτόν. Στρέφομαι και προς τους ε, δύο. Όχι, προ του τρει. Ο κύριο Ντελάνο, ο κύριο Ντεπρέ συμφωνούν. Ο κύριο Γκάιερ που επανήλθε συμφωνεί. Ωραία, σα ευχαριστώ κύριε. Διάφορα, αν δεν υπάρχουν, λήξη τη συνεδρίαση θα τα πούμε αύριο στι 9. Όπου έχουμε ψηφοφορίες.